και η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ήδη μελετούν το προσχέδιο μέτρων της ε, κυβέρνησης προκειμένου να δει ποια θα είναι τα βήματα που θα αναλάβει στο μέλλον η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όλες οι εναλλακτικέ λύσεις προφανώς προς το παρόν και τα διαβήματα είναι ανοιχτά. Ε, Uh, uh, Σε ό,τι αφορά την έκθεση Howitt, θα ακούσουμε πρώτα τον εισηγητή, τον κύριο Howitt και μετά. Ε, είχε ε, προβλεφθεί να μιλήσει πρώτα η κυρία Άστον, αλλά κάνουμε μια μικρή αλλαγή και δίνουμε το λόγο στον εισηγητή, τον κύριο Howitt. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Η συζήτησή μα για την ατήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα έρχεται σε μια σημαντική στιγμή γιατί μα επιτρέπει να ε, συμβάλλουμε στην στρατηγική ε, ανασκόπηση ε, και να προτείνουμε τα θέματα που είναι πολύ σημαντικά για μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όταν απειλούνται τα ανθρώπινα δικαιώματα, η έκθεση αυτή πρέπει να το επισημάνει. Ε, επίσης, ε, αναφερόμαστε στον θυνατότητα ε, διορισμού ενός ειδικού εκπροσώπου για τα ανθρώπινα δικαιώματα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να βρίσκονται τα ανθρώπινα δικαιώματα σε ίδια μοίρα στο Συμβούλιο με άλλα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Θα ζητάμε ένα χρονοδιάγραμμα βάσει του οποίου θα εργάζονται οι αντιπροσωπείε μας σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα σε ολόκληρο τον κόσμο και ζητούμε η κοινωνία των πολιτών και οι οργανώσεις τη να αντιμετωπίζονται ω ίσοι εταίροι. Όταν υπάρχουν ε, ε, ε, οι εικασίε για παραβιάσει των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να παραβλέπουμε αυτά που γίνονται εκτό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να αυξηθεί σε τεράστιο βαθμό η διαφάνεια όσον αφορά την πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, διότι ε, οι στόχοι μα όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα μπορούν να επιδηθούν μόνο όταν υπάρχει λογοδοσία. Αναφέρουμε εδώ έξι χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν έχουν επικυρώσει τα σχετικά με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Επίσης υπάρχουν 13 χώρες που ούτε, είτε δεν υπέγραψαν είτε δεν επικύρωσαν το πρωτόκολλο των Ηνωμένων Εθνών κατά των βασανιστήριων. Και για να φέρω τη δική μου χώρα, το Ηνωμένο Βασίλειο, το οποίο ε, παρεμπόδισε την επικύρωση ε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση της ε, Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Προς την ε, είπατε εκπρόσωπο, ήθελα να πω ότι καταλαβαίνω το δόγμα περισσότερο για περισσότερο όσον αφορά την αραβική ε, άνοιξη. Ε, να σκεφτούμε όμως τι έγινε με τον Καντάφη ε, τέσσερις εβδομάδες πριν αρχίσουμε να τον βομβαρδίζουμε. Ίσως τώρα θα πρέπει να μιλάμε για λιγότερα για λιγότερα. Οι διεθνείς συμφωνίες δεν χρησιμοποιούνται αποτελεσματικά. Ζητούμε κριτήρια και benchmarks για κάθε χώρα και μηχανισμούς που θα επιτρέπουν πραγματικά μια κλιμάκωση στις αντιδράσεις. Πρόεδρε, έχω υποστηρίξει ότι, ότι η υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι πιο ε, σημαντικό θέμα ε, από όλα. Και γι' αυτό θα έπρεπε να ε, συγχαρούμε το Βέλγιο και την Αυστρία που ε, υιοθέτησαν προτάσεις για τις ε, και για την Γάζα. Ε, επίσης καλωσορίζουμε την ε, συνεργασία των ε, σκιωδών εισηγητών για θέματα που δεν είναι πάντοτε πάρα πολύ εύκολα. Είχε διαρθεί η Επιτροπή για θέματα ισότητας των γυναικών για έκτακτες παραδόσεις κλπ. Στην έκθεση αυτή ε, ιδιαίτερα αναφέρομαι στο θέμα των κοινωνικών ε, μέσων επικοινωνίας και των επιχειρήσεων σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Υπάρχει συνεχής αύξηση των χρήσεων των νέων τεχνολογιών. Υπάρχει όμως παράλληλα μια χαλιναγώγηση των μέσων ε, αυτών και αυτών που τα χρησιμοποιούν με σκοπό την απελευθέρωση. Ε, ε, αν σκεφτούμε τι έγινε με το Μουμπάρακ ή ε, με το Google ε, που δεν υπέκυψε στις πιέσεις της Κίνας. και αργότερα θα επανέλθουμε στο θέμα της εταιρικής ευθύνης στο σημείο αυτό. Επίσης, η Ευρώπη θα πρέπει να βρεθεί σε ίση μοίρα με το ε, με, τα, με τις ΗΠΑ που έχουν έναν ε, υπουργό για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πρέπει και εμείς να αποκτήσουμε έναν ε, το εκπρόσωπο για τα ανθρώπινα δικαιώματα. πρέπει να δείξουμε ότι καταλάβαμε όλα τα διδάγματα που υπήρχαν και πριν από την Αραβική Άνοιξη. Η ελευθερία έκφρασης έχει ένα νέο νόημα σε αυτό τον κόσμο που δημιουργείται. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε συνάδελφε Χάουιτ. Ο κύριος Πρέντα από την Επιτροπή Ανάπτυξης. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είμαι ο συντάκτης της γνωμοδότησης της Επιτροπής Ανάπτυξης για το θέμα αυτό και θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Χάουιτ και να τον ευχαριστήσω για τη συμπερίληψη του συνόλου σχεδόν των παρατηρήσεών μας στην τελική του έκθεση. Είμαστε υπέρ μιας αποτελεσματική συμπερίληψη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην αναπτυξιακή βοήθεια, κάτι που ανταποκρίνεται και στη λογική τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Και η νέα προσέγγιση σε ό,τι αφορά την λήψη υπόψη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη δημοκρατία είναι ευπρόσδεκτη και ε, κατοχυρώνει μια ολοκληρωμένη στρατηγική των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που καλύπτει όλε τι πτυχέ των κοινοτικών πολιτικών. Βέβαια θα πρέπει για να περάσουμε από τα λόγια στα έργα να διανύσουμε πολύ σημαντικό δρόμο και η δημοσιονομική στήριξη θα πρέπει να εξαρτάται από την κατάσταση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και χρηστής διακυβέρνηση στις χώρες δικαιούχους. Και όλα αυτά θα πρέπει να τα εξηγήσουμε με πολλές λεπτομέρειες. Είναι δύσκολο βέβαια να μιλούμε για, ε, σε περίοδο οικονομικής κρίσης για αύξηση του προϋπολογισμού, αλλά θα πρέπει να ενισχύσουμε την πρικοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Δημοκρατίας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, γιατί ε, έτσι θα προάγουμε και με αυτό τρόπο τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστώ από την Επιτροπή για τα δικαιώματα της γυναίκας. Ο κύριος Ιμένες για ένα λεπτό παρακαλώ. Η κυρία. Η κυρία Ιμένες δεν είναι στην ε, ε, αίθουσα. Δίνω λοιπόν το λόγο στην ε, Αντιπρόεδρο κυρία Άστον. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Από το 1983, όταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπήκε στη διαδικασία έγκρισης της ετήσιας έκθεσης και του ψηφίσματος για τα ανθρώπινα δικαιώματα, το Κοινοβούλιο αυτό έκανε περισσότερα πράγματα από κάθε άλλο θεσμικό όργανο για να επικεντρωθεί στο θέμα. Μπορεί καμιά φορά να διαφωνούμε σχετικά με το πώς θα προβάλλουμε και θα στηρίξουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα και το σεβασμό του σε όλο τον κόσμο. Είμαστε ενωμένοι στο στόχο μα να δημιουργήσουμε ένα πιο ελεύθερο κόσμο όπου θα γίνει, την χάνει σεβασμού η ανθρώπινη αξιοπρέπεια ε, όπου και, από όπου και αν προέρχονται οι άνθρωποι αυτοί και ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης ειδικότερα ε, ο σκοπός είναι να παίξουν έναν ρόλο πολύ σημαντικό στην υποστήριξη του αγώνα των ανθρώπων για τα δικαιώματά τους. Περνώ τώρα στην έκθεση του κυρίου Χάουιτ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το κείμενο αυτό και για μένα και για τους συναδέλφους στην Επιτροπή και το Συμβούλιο. Ήδη η πρώτη πρώτη παράγραφος ε, στην έκθεση Χάουιτ αφορά τη συνοχή μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα από τα βασικά θέματα της ε, ανακοίνωσης του Δεκεμβρίου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα για το Κοινοβούλιο αυτή την εβδομάδα, επειδή την Πέμπτη θα ακούσετε δηλώσεις από το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Η λέξη συνοχή μπορεί να ακούγεται ξερή λέξη, αλλά σημαίνει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα θα εντάσσονται σε οτιδήποτε κάνουμε στην Ευρώπη και εκτός Ευρώπης. Σημαίνει ότι θα διασφαλίζομαι ότι οι άνθρωποι παντού θα ωφελούνται από τα ίδια καθολικά οικουμενικά δικαιώματα, ανεξάρτητα από το ποιοι είναι και που ζουν. Θα ήθελα να αναδείξω δύο θέματα. Ε, καταρχήν την ε, λογοδοσία και τη σημασία της και τη σημασία του έργου μας ε, σχετικά με το πώς αναπτύσσουμε τη λογοδοσία σε σοβαρές καταστάσεις. Επικεντρώνουμε σε δύο θέματα τα οποία αφορούν την συνοχή και τη λογοδοσία. Ε, στο ρόλο των γυναικών, είδα την Μισελ Μπασουλέ για να μιλήσω για το ρόλο των γυναικών και ε, για το πώς θα προχωρήσουμε και μαζί με τα Ηνωμένα Έθνη για να στηρίξουμε τις γυναίκες σε όλο τον κόσμο. Και η ε, διακρίσεις κατά των χριστιανών, ε, ανθρώπων που δεν έχουν συγκεκριμένη πίστη ή άλλων ε, ομάδων θρησκευτικών εντείνονται γι' αυτό. Θα πρέπει να ενισχύσουμε την πολιτική μας για την ελευθερία θρησκείας ή πίστης που είναι πολύ σημαντική σε μια ελεύθερη κοινωνία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να ε, υπάρχει ε, ένας ε, κανονισμός που και το καταστατικό της Ρώμης υπάρχει πρόοδος εδώ και ήδη έχουν υπογραφεί τρεις διμερείς συμφωνίες. Έχουν μονογραφεί τρεις ακόμη και γίνονται διαπραγματεύσεις για 15. Εμείς έχουμε την δυνατότητα να προωθήσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα Ε, τοποθετώντας ε, χώρες και καθεστώτα ε, σε ένα φάσμα το οποίο καλύπτει διαφορετικές καταστάσεις από την απομόνωση μέχρι την πλήρη ένταξη. Τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν ήταν ποτέ σημαντικότερα και ποτέ δεν έχουν υποστεί τόσες αλλαγές. Ε, μπορούμε να πάρουμε παραδείγματα από τη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική, όπου νέοι, ηλικιωμένοι, άνδρες, γυναίκες, εκπρόσωποι όλων των κοινωνικών στρώματων, ε, πάλεψαν, πολλοί θυσίασαν και τη ζωή τους για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ελευθερία, την αξιοπρέπεια, ένα καλύτερο μέλλον. Θα ήθελα να αποτίσω φόρο τιμής σε όλους αυτούς εδώ. Οι αλλαγές που επέφεραν, όπως είπε και ο κύριος Χάουιτ, ε, απαιτούν και από την Ευρωπαϊκή Ένωση κάποιες ε, ε, αλλαγές. Ανταποκριθήκαμε στην πρόκληση με τα ανθρώπινα δικαιώματα και η πολιτική μας προς τους γείτονες τώρα έχει γίνει ισχυρότερη και πιο υγιής ως αποτέλεσμα. Επίσης έγινε προσπάθεια για να ενισχυθούν οι θετικές εξελίξεις. Ε, στην 19η Σύνοδο ε, ε, το ψήφισμα για την Συρία εγκρίθηκε με 41 από 47 ψήφους επίσης και το ψήφισμα για την βερμανια Μιανμάρ έγινε δεκτό ε, επίσης ε, ήταν πολύ σημαντική η σύνοδος αυτή για τα δικαιώματα ε, ατόμων που πολλές φορές περιθωριοποιούνται ή εξωστρακίζονται. Βία, εγκλήματα φύλου αντιμετωπίστηκαν επιτυχώς και με την υποστήριξη του Μπανκιμούν. Δεν είναι, είναι απαράδεκτο 80 κράτη ακόμα να ποινικοποιούν στις ίδιες στις σεξουαλικές σχέσεις μεταξύ ε, ενηλίκων ε, που συμφωνούν ε, είναι, ήταν πολύ σημαντικό το γεγονός ότι οι σύνεδροι μπόρεσαν να ασχοληθούν ε, με ε, όλα αυτά τα θέματα ε, και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πραγματικά αναδείχθηκε ως θεσμικό όργανο το οποίο προωθεί τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο. Η ανακοίνωσή μου του περασμένου Δεκεμβρίου ήταν μια συμβολή στη συνεχιζόμενη συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για πιο αποτελεσματική και συνολική προσέγγιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της ε, δημοκρατίας. Τώρα ε, έχετε εξετάσει τις προτάσεις. Ε, όπως επιβεβαίωσα στην άφετη στις 20 Μαρτίου, τώρα γίνονται εργασίες για να προχωρήσουμε το ζήτημα του διορισμού ειδικού εκπροσώπου για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι σημαντικό το πρόσωπο αυτό είναι κάποιος με ε, λαμπρά επιτεύγματα στα θέματα ε, διεθνών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Επίσης, ε, όπως συζητήθηκε στην συνάντηση στο Κίμνιχ, θα συμφωνήσω για ε, μία, πάνω σε μια πολιτική δήλωση σχετικά με τους στόχους μας. Αυτό θα ε, συγκεράσει πολλές νέες πρωτοβουλίες. Χαίρομαι διότι επιβεβαιώνω ότι το Δίκτυο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των ε, Σημείων Εστίασης ήδη έχει ολοκληρωθεί αφού 116 αντιπροσωπείες Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν ένα σημείο επαφής, ορισμένες έχουν δύο. Ε, θα ήθελα σε αυτά τα, πάνω σε όλα αυτά τα θέματα να συνεργαστώ στενά μαζί σας. Η ε, επανεξέταση και αναθεώρηση της πολιτικής ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Ένωσης πρώτη φορά ανακοινώθηκε σε αυτό το κοινοβούλιο. Ο διορισμός ειδικού ε, προσώπου ε, βρήκε το κοινοβούλιο σύμφωνο. Απευθυνά επιστολή στον πρόεδρο της Επιτροπής ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, για και στην κυρία Μπάρβαλα Λοχμπίλντερ, ούτως ώστε να συνεργαστούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ευχαριστώ τον κύριο Χάουιτ για την έκθεση και συγχαίρω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για το συνεχιζόμενο έργο του στον τομέα της προώθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ευχαριστώ κυρία Αντιπρόεδρε. Το λόγο τώρα έχουν οι ομιλητές εκ μέρους των πολιτικών ομάδων. Ο κύριος για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η φετινή έκθεση έπρεπε ήδη να έχει εγκριθεί από το Δεκέμβριο του 2011. Είμαστε όμως ήδη στο πρώτο τετράμινο του 2012. Βέβαια, εξετάζουμε αυτή την έκθεση σε συνδυασμό με την Ευρωπαϊκή Πολιτική για τον Εκδημοκρατισμό και τα ανθρώπινα δικαιώματα μετά την ανακοίνωση που υπέβαλε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η ύπατη εκπρόσωπος τον προηγούμενο Δεκέμβριο. Πολλά συνέβησαν στα ανθρώπινα δικαιώματα το 2010. Βέβαια, λαμβάνοντας την έκθεση αυτή αναχήρας, δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τις εντυπώσεις που μας άφησε η αραβική έκθεση και που τροποποιεί την προσέγγιση μας στα θέματα εκδημοκρατισμού και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μια νέα προσέγγιση για τα θέματα αυτά ε, θα πρέπει να περιλαμβάνει τη συνέργεια μετά την εμπειρία από την Αραβική Άνοιξη και φυσικά την ε, ευθυγράμμισή μας με τις νέες διατάξεις της συνθήκης ε, της Λισαβόνας. Με ιδιαίτερη ικανοποίηση δέχομαι την έκθεση του κυρίου Χόουιτ. Τον ευχαριστώ θερμά για την αγαστή συνεργασία που, είχαμε, με το, που είχε ο εισηγητής με το ΕΛΚ. Βέβαια αναφέρονται κάποιες επικρίσεις στη Λευκορωσία για την καταστράτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναφέρθηκε ε, παραβίαση των δικαιωμάτων των κρατουμένων, ε, την εφαρμογή της, ε, την, την εσχάτη των ποινών που εξακολουθεί να ισχύει ακόμη, την στέρηση πληροφορίας των συγγενών των καταδικασμένων και γενικώ ε, περιορισμό των δικαιωμάτων. Συμφωνώ με την έκκληση για την επιφυλάκηση των δύο πολιτικών κρατουμένων. Και έχουμε και το πρόσφατο ψήφισμα του Euronest στον Πακού σε ό,τι αφορά την ε, συμμόρφωση των ε, χωρών της γειτονίας σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και χαίρομαι ιδιαίτερα για τη μνήα της, του, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Δημοκρατίας που θα υποστηρίξει τον εκδημοκρατισμό και την μεταρρύθμιση και τις δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις στις διάφορες χώρες. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη, να λάβουμε υπόψη και τα δικαιώματα των θρησκευτικών κοινοτήτων, ιδιαίτερα των χριστιανών. Δεν μπορούμε να δεχτούμε διώξει ούτε χριστιανών ούτε ένα άλλο θρησκευτικών κοινοτήτων. Και φυσικά είναι σημαντικό ο ρόλο τη πρωτοβουλία ε, και των συνηγόρων των πολιτών και αναφέρθηκε ιδιαίτερα η συνεργασία του Γάλλου και του Πολωνού συνηγόρου του πολίτη. Νομίζω ότι είναι σημαντική αυτή η ανταλλαγή των βέλτιστων πρακτικών και θα στηρίξουμε έτσι τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τέλος, θα ήθελα να αναφερθούμε και στην εταιρική ευθύνη. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τι εμπορικέ μα σχέσει με γειτονικέ χώρε Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά. σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Κοπά για δύο λεπτά, εκ μέρους των συλληστών. Να συγχαρώ τον συνάδελφο Ρίτσαρντ Χάουετ για την περιεκτική και ιδιαίτερα εμπεριστατωμένη έκθεσή του, αλλά και την ε, ύπατη εκπρόσωπο λέιδι Άστον για τη σταθερή προσήλωσή της στα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι αναγκαίο πλέον να λάβουμε τα μηνύματα των καιρών και να κάνουμε την αυτοκριτική μας. Να δείξουμε ότι μάθαμε από τα λάθη μας δυστυχώς η δύση και τα κράτη μέλη της ευρωπαϊκής ένωσης για χρόνια υποστήριξαν ενεργά ή παθητικά τα δικτατορικά καθεστώτα της βόρειας αφρικής στο όνομα μιας επίπλασης σταθερότητας. σήμερα είναι πλέον σαφές και όλοι μας νομίζω αντιλαμβανόμαστε ότι δεν μπορεί να υπάρχει μακροχρόνια σταθερότητα χωρίς σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία. εφόσον θέλουμε πραγματικά να είναι η ευρωπαϊκή ένωση αξιόπιστος δρόν στο διεθνές στερέωμα πρέπει επιτέλους να αποφευχθούν οι πρακτικές δύο μέτρων και δύο σταθμών στο ζήτημα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. κάθε είδους βοήθεια που προσφέρεται σε τρίτες χώρες πρέπει να συνοδεύεται από αποτελεσματική πίεση για έμπρακτες βελτιώσεις στον τομέα αυτό. σε αυτό το πλαίσιο η ρήτρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις εμπορικές συμφωνίες που συνάπτει η ένωση με τρίτες χώρες είναι ένα σημαντικό εργαλείο που πρέπει κατάλληλα να αξιοποιηθεί. και γενικά πρέπει να είναι σαφές ότι η λογική του more for more συνεπάγεται και το less for less. είναι επίσης σημαντικό τα κράτη μέλη να μιλάνε με μια φωνή στον οργανισμό ηνωμένων εθνών και σε άλλα σημαντικά διεθνή φόρα. καλωσορίζουμε λοιπόν την υιοθέτηση των γενικών κατευθύνσεων σχετικά με τις δηλώσεις της ευρωπαϊκής ένωσης στα διεθνή φόρα. επαναλαμβάνουμε όμως παράλληλα την έκκλησή μας για τακτικές διαβουλεύσεις μεταξύ των πρέσβεων των κρατών μελών της ένωσης προκειμένου να επιτευχθεί καλύτερος συντονισμός στην κοινή προσπάθεια για την προώθηση και προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. δύο σημεία τέλος. πρώτα απ' όλα η ανάγκη να υπερασπιστούμε την θρησκευτική ελευθερία είναι αυταπόδεικτη. πρέπει όμως να αγωνιστούμε για την ελευθερία όλων ανεξαιρέτως των θρησκευτικών ομάδων και όχι μόνο των χριστιανικών όπως ζητούν κάποιες ομάδες σε αυτό το κοινοβούλιο και τέλος θέλω να σταθώ στο θέμα των αναπαραγωγικών δικαιωμάτων των γυναικών. το δικαίωμα στο σώμα για κάθε γυναίκα είναι ένα βαθιά ανθρώπινο δικαίωμα δικαίωμα στην αξιοπρέπεια και την ελευθερία. για όλους εμάς που η ελευθερία είναι ένα αδιαπραγμάτευτο δικαίωμα το δικαίωμα κάθε γυναίκα στο σώμα της είναι κεντρικό. σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την ομάδα Άλντε. Ο κύριος Ντόνσκης για δύο λεπτά. Thank Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να συγχαρώ τον συνάδελφο, τον κύριο Χόουιτ, για την καταπληκτική του έκθεση, γιατί θεωρώ ότι η επανασυμφιλίωση των πολιτικών και των ε, ε, ηθικών ευαισθησιών της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης και των πολιτικών είναι σημαντική πρόκληση. Η έκθεση διαρωτάται πότε τα ανθρώπινα δικαιώματα βρέθηκαν στο επίκεντρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση και θα συμπεριληφθούν οριζόντια σε όλε τι πολιτικέ και θα αποτελέσουν ακρογωνιαίο λίθο και τη εξωτερική πολιτική. Επίση, πότε έγιναν τα ανθρώπινα δικαιώματα κοινό παρανομπαστής από πολιτική και ηθική άποψη σε όλε τι πολιτικέ παρατάξεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι σε ό,τι αφορά κατάφορε παραβιάσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπω είναι δολοφονίες, ε, ε, θανατική καταδίκη, παραβίαση των ελευθεριών έκφρασης, πολιτικών επιθυμι... Ε, επιθύσεων, η δίωξη των ομοφυλοφίλων, υπάρχουν κάποιες κοινέ αρχές, γιατί είναι κοινέ αυτές οι αξίες μας και η συμπεριφορά μας. Πάντως πιστεύω ότι η πρόκληση του μέλλοντος έγκυται στην ικανότητά μας να εντοπίσουμε και να αντιμετωπίσουμε λιγότερο κατάφορες, πολύ πιο διακριτικές και λεπτές ε, ε, παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως επιλεκτικές πολιτικοποιημένες δίκες, εκφοβισμό, που ε, υπονομεύει την ίση μεταχείριση, κατάχρηση της ψυχιατρικής, ε, εκβιασμό και άλλες μεθόδους εκφοβισμού ε, ακτιβιστών ή ιδιωτών. Νομίζω πάντως ότι σε κάθε περίπτωση ο εισηγητής μας στο μέτρο των δυνατοτήτων του επιτέλεσε εξαιρετικό έργο και πιστεύω ότι η έκθεση καλύπτει ένα τεράστιο πεδίο των ευαισθησιών, των μελημάτων μας και των προσδοκιών μας και για όλες αυτές τις προσπάθειες συγχαίρω θερμά τον εισηγητή μας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τους πράσινους. Ο κύριος Ταβάρης για 1,5 λεπτό. Σας ευχαριστώ. Κυρία ε, Άστον, ομολογώ ότι έμεινα ευρώντητος από τη δρόμη σας έμεινε βρόντιτος από την, την πρώτη σας ε, παρέμβαση για τη διαδικασία απαλωτρίωσης της Ρέψολ από την κυβέρνηση της ε, Αργεντινή. σε μία συζήτηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, και έχοντα υπόψη τη μία από τι χώρε που χρησιμοποιήθηκαν ω πλατφόρμα για τη λαθρεμπόριο όπλων, το μόνο που κάνατε ήταν ένα απλό ανακοινωθέν τύπου. Ενώ ε, σε μια χώρα από την οποία αποσύραμε την ε, αντιπροσωπεία μας και δεν την έχουμε αποκαταστήσει, σε μια χώρα της Δυτικής Αφρικής που θα μετατραπεί σε άναρχο κράτος, αν δεν έχει ήδη μετατραπεί, Εκεί δεν μας είπατε τίποτα. Μακάρι και για τις δύο αυτές περιπτώσεις να είχατε δράσει τόσο άμεσα όπως και κάνατε και με την περίπτωση Ρεψόλ. Έχουμε ε, παράνομη εισαγωγή, λαθρεμπόριο ε, όπλων στη Συρία. Υποστηρίζουμε έμεσα δικτατορικά καθεστώτα, ενώ έχουμε και αποφάσεις διεθνείς χωρίς ε, καμία μνήμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Σπεύσατε ε, να προστατεύσετε βέβαια τις επιχειρήσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, αλλά φαίνεται ότι δεν ενδιαφέρει τόσο για τα ανθρώπινα δικαιώματα. έχουμε κοινέ στρατηγικές, κρατικές στρατηγικές και εναρμόνιση των εσωτερικών και των εξωτερικών πτυχών τη πολιτική για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστώ τον κύριο Χάουιτ και για την συνεργασία και για τι πολύ ε, έμπρακτε προτάσει τη έκθεσή του και εύχριστε. Πιστεύω ότι η έκθεση αυτή είναι πολύ χρήσιμη και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και ω κοιόδη ε, εισηγητή τη έκθεση Χάουιτ, και συνεισηγητή για την αναθεώρηση τη θετική ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων τη Ευρωπαϊκή Ένωση, πιστεύω ότι ήρθε η ώρα να τελειώσουν οι φάρσε, να αφήσουμε τα αστεία και να ξεκινήσουμε ένα πολύ πιο σοβαρό έργο για τα ανθρώπινα δικαιώματα, κυρία Άστον. Ε, Ευχαριστώ για την ομάδα των ε, ε, συντηρητικών και μεταρρυθμιστών, ο κύριος Σιμάνσκι, για δύο λεπτά. Κυρία, είπατε εκπρόσωπε, κυρίες και κύριοι. Η φετινή έκθεση για τα θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο σε μερικές περιπτώσεις αποτελεί σημαντική πρόοδο σε σχέση με προηγούμενα κείμενα, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την ανεξιθρησκεία. Η θρησκευτική ελευθερία αποτελεί αναπαλωτήριο το τμήμα των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ο θεμελιώδης χαρακτήρας ε, επιβεβαιώνεται και στη Συμβάση του ΟΗΕ και του Συμβουλίου της Ευρώπης. Μάλιστα η αυξανόμενη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ιδιαίτερα των χριστιανών, αποτελεί σημαντική αύξηση των ε, παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο. Και μια χρονιά που μετά την έναρξη της ε, ε, Αραβικής Άνοιξης υπάρχουν σοβαρές απειλές για ολόκληρη την χριστιανική κοινότητα στην Αγγής Ανατολή. Θα ήταν πραγματικά τραγικό αν διαπιστωθεί ότι οι χριστιανοί θα είναι τα πρώτα θύματα αυτής της πολυπόθητης ε, δημοκρατίας και του εκδημοκρατισμού στην Αγγλική Ανατολή. Θα πρέπει αυτό να το υποθυμίζουμε στους πολιτικούς μας εταίρους. Δύσκολα συμφωνήσουμε με τις επικρίσεις κατά της ε, Γαλλίας και της Μεγάλης Βρετανίας ό,τι αφορά την πολιτική τους ε, για το πρόβλημα της προσχώρησης Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Γιατί κάτι τέτοιο ε, ίσως δημιουργήσει ε, σύγκρουση δικαιοδοσιών μεταξύ δικαστηρίων του Λουξεμβούργου και του Στρασβούργου και να δημιουργήσει ανεξέλεκτη αύξηση των αρμοδιοτήτων των κοινοτικών δικαστηρίων. Ε, πιστεύω ότι από την έκθεση θα πρέπει να αφαιρεθούν κάποιε αναφορέ στην απαραγωγική υγεία, γιατί τέτοιου είδου διατάξει αποτελούν πρόσχημα στην προαγωγή και τη χρηματοδότηση των αυλώσεων στον κόσμο. Και μάλιστα ακόμη και σε χώρες που θεωρούν ω αξιόπινες τι ε, αμβλώσεις. Κάτι τέτοιο συνιστά τεράστια κατάχρηση τη εμπιστοσύνη των πολιτών και των κρατών μελών που ουδέποτε δεν ανέθεσαν τέτοιου είδου αρμοδιότητε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ για την ομάδα ε, Ευθερίας και Δημοκρατίας. Ο κύριος Πέλτε για δύο λεφτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, τα τελευταία χρόνια, στι τελευταίε μέρε στην Ολλανδική τηλεόραση, είδαμε κάποια συγκλονιστικά ρεπορτάζ και εικόνε ε, σε ό,τι αφορά απαγωγέ και εξαναγκαστικούς προσυνετελισμούς στο Ισλάμ νεαρών γυναικών και κοριτσιών ε, χριστιανών στην Αίγυπτο. Και μάλιστα είδαμε οι των σταυρών που τους, τους έσπαζαν μπροστά στις γυναίκες αυτές που έτρεχαν απεγνωσμένα προκειμένου να γλιτώσουν από τους δημίους τους. Ήδη το Δεκέμβριο του 2011, κυρία είπατε εκπρόσωπε, απαντήσατε σε ερωτήσεις μας για τις σοβαρές κατάφορες παραβιώσεις των δικαιωμάτων αυτών των θρησκευτικών χριστιανικών μειονοτήτων στην Αίγυπτο και μιλήσαμε για, τις, ε, για τους προβληματισμούς μας ό,τι αφορά τις απαγωγές και τις, τους εξαναγκαστικούς προσιλητισμούς. Μάλιστα στείλαμε και επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκειμένου να συμβάλλουμε και εμείς στην ε, ε, λήψη κάποιων μέτρων αυτής της εξοργιστικής κατάστασης. Ήταν συγκλονιστικές εικόνες στην τηλεόραση και κάποιες εκκλήσεις της Εκκλησίας να σταματήσει μια τέτοια πρακτική. Μάλιστα είχαμε από τις παλιότερες οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αίγυπτο που μας είπε ότι τα, τους τελευταίους μήνες 1500 γονείς κατήγγυλαν απαγωγές των παιδιών τους, κυρίως των κοριτσιών τους. Οι περισσότερες ε, ήταν ανήλικες μάλιστα και μόνο 10 τέτοια κόρης έχουν ξαναβρεθεί, 10 τέτοιες απαγωγές έχουν διαλευκανθεί. Μάλιστα είδαμε τις εικόνες ενός ε, ζευγαριού από την Αίγυπτο που έβλεπε ε, στην τηλεόραση την ε, κόρη τους 15 ε, ετών που με κλάματα, με δάκρυα στα μάτια ζητούσε από τους γονείς ε, να προσχωρήσουν στο Ισλάμ, να προσιλητιστούν αν ήθελαν να την ξαναδούν ζωντανή. Νομίζω ότι θα πρέπει να αναλάβουμε κάποια διαβήματα απέναντι στις Αιγυπτιακές αρχές, να προσκαλέσουμε τις Αιγυπτιακές αρχές να διαλευκάνουν τις περιπτώσεις αυτές, να λάμψει η αλήθεια και να αποκατασταθεί ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων αυτών, των, αυτής της πολύ σημαντικής θρησκευτικής μειονότητας που είναι χριστιανοί της Αιγύπτου. Παρακαλώ, κυρία Πρόεδρε, κυρία Υπατή Πρόσωπο, να δώσουμε συνέχεια σε αυτά τα περιστατικά και να μας ενημερώνετε. Εκ μέρους της Γκουέ, κυρία Βεριζιά, για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τον εισηγητή μας, τον Ρίτσαρτ Χόουιτ, γιατί πραγματικά Ποτέ δεν είχα προηγουμένω την ευκαιρία να εργαστώ σε ένα τέτοιο ε, κλίμα και ποτέ δεν είδα έναν ε, εισηγητή να είναι τόσο πρόθυμος ε, για συνεργασία και για συμβιβασμούς. Μερικές φορές προσπάθησε να συμβάσει και τα συμβίβαστα. Σίγουρα θέλουμε να σημειώσουμε πρόοδο ότι αφορά τι απαιτήσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ιδιαίτερα τη Ευρωπαϊκή Ένωση για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η έκθεση επιμένει στην ανάγκη συνδυασμού της εξωτερικής και εσωτερικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυτό. Και εκεί πολύ δρόμο έχουμε να διανύσουμε, γιατί πριν να κάνουμε κηρύγματα και να δίνουμε μαθήματα σε όλο τον κόσμο, θα πρέπει πρώτα να διορθώσουμε τα του οίκου μας και δυστυχώς πολλές φορές διαπιστώνουμε υποκρισία στην περίπτωση αυτή. Η έκθεση επιμένει στην ανάγκη έμπρακτης εφαρμογής των ρητρών δημοκρατία και ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι ρήτρε αυτέ δεν θα πρέπει να βρίσκονται μόνο για να καθησυχάσουν τη συνείδησή μα, γιατί θα είναι τελείως άχρηστες αν, στις, αν συνεχώς θυσιάζονται στο βωμό του οικονομικού φιλελευθερισμού. Θα πρέπει να εφαρμόζουμε εμπράκτως τις ρήτρες αυτές. Δεν συμφωνώ με τα θετικά σχόλια ε, ως το πρόσωπό σας για την πολιτική γειτονία. Ε, λυπούμε, αλλά διαφωνώ με τις θετικές αυτές παρατηρήσεις. Τι γίνεται σε ό,τι αφορά το Ίδρυμα για την υποστήριξη της δημοκρατίας. Υπάρχει κίνδυνος πολιτικής χειραγώγησης με μια κακή χρήση αυτού του μέσου. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ για τους μη ε, γεγραμμένους Ο κύριος Κλάης για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να επισέλθουμε σε όλες τις λεπτομέρειες των εκθέσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εγώ θα αναφερθώ όμως σε κάτι που δεν αναφέρθηκε στην έκθεση. Ε, η κατάσταση στην Νότια Αφρική και ιδιαίτερα τους λευκούς ε, αγρότες. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα εγκληματικότητας, ε, όλες οι εθνωτικές ομάδες πλήττονται, αλλά η συστηματική επίθεση κατά των λευκών αγροτών είναι σαφής και πρέπει να προσεχθεί από εμάς. Τα τελευταία 15 χρόνια δολοφονήθηκαν περίπου 3.000 κάτω από άγριες συνθήκες. Ακόμα και παιδιά ε, σφαγιάστηκαν. Είναι μια πολύ ευάλωτη ομάδα αυτή, μια μικρή μειονότητα και επίσης λόγω της γεωγραφικής ε, κατανομής τους πολλά αγροκτήματα είναι σε απομακρυσμένες περιοχές. Το παρατηρητήριο γενοκτονίας των Ηνωμένων Εθνών ε, και το Αμερικανικό Παρατηρητήριο έχει επιστήσει την προσοχή σε αυτό το θέμα και μίλησαν για γενοκτονία. Πολλά εγκλήματα γίνονται στη Νότια Αφρική. Υπάρχει συστηματική εκστρατεία κατά των αγροτών αυτών και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να κάνουμε τα πάντα για να αποφύγουμε περαιτέρω κλιμάκωση της βίας. Φεύγουν όλο και περισσότεροι αγρότες από την Νότια Αφρική και στο τέλος η κατάσταση θα γίνει όπως στο Ζιμπάμπουε. Θα πρέπει να ε, μπει ένα τέλος σε αυτή την κατάσταση και απευθύνω έκκληση δηλαδή Άστο να καταδικάσει στεναρά τη βία κατά των αγροτών και να αναστείλει την βοήθεια στην Νότια Αφρική αν δεν ληφθούν αποτελεσματικά μέτρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Το λόγο έχουν τώρα οι άλλοι ομιλητέ, ξεκινώντας με τον κύριο Σαλαφράγκα για δύο λεπτά. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Υπουργέ κυρίες και έκθεση του κυρίου Χόουιτ ε, αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα που είναι πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά. Γι' αυτό, κυρία Άστον, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω ιδιαίτερω για την ε, δήλωσή σα πριν την άνοιξη συζήτηση επί της έκθεση Χάουιτ για την κατάσταση στην επιχείρηση Ρεψόλ. Δεν, είπατε, δεν θα μπορούσατε σε τόσο λίγο χρόνο να, πείτε, να κάνετε και να πείτε τόσο περισσότερα. Λάθος απόφαση, απειλή για τις ε, αλλοδαπές επενδύσεις στη χώρα αυτή, ανάγκη να ε, τηρηθούν οι λιμένες δεσμεύσεις και υποχρεώσεις. Τα, το γεγονό ότι συμπεριληφθήκε στην ημερήσια διάταξη του ε, Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών και την ε, αναστολή, αναβολή μάλλον της ε, Μεικτής Επιτροπής Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, Αργεντινής όσο του ε, ληφθούν κάποια μέτρα. Η έκθεση Howitt είναι λογική, βέβαια εκκρεμούν κάποιες ε, υποθέσεις, κάποια ζητήματα όπως η αποστολή της ερευνητικής των πραγμάτων αποστολής στη Γάζα ήταν ένα είναι ένα αίτημα που δεν μπορούμε να δεχτούμε στην ομάδα, όπως ξέρετε. Και η θέση σας για την Κολομβία, κύριε Χόουιτ, ε, είναι παραλυρηματική κατά κάποιο τρόπο. Γι' αυτό απορρίψαμε το σχετικό σημείο στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και μάλιστα ενώ περιμένουμε την ε, κύρωση της ε, πολυμερούς συμφωνίας με την Κολομβία δεν είναι δόκιμα τα σχόλιά σας για τη χώρα αυτή. Θα ήθελα να αναφερθώ, κυρία Άστον, σε ένα θεμελιώδες ε, θέμα της πολιτικής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που είναι προσφυλές ε, για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το θέμα του διορισμού του ειδικού εντεταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η πατορμοστή για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα αποφανθούμε για το θέμα αυτό σε ένα ψήφισμά μας ε, και θα ήθελα η διαδικασία και η εκλογή του προσώπου αυτού να είναι αντικειμενική και πραγματικά να αναλάβει το έργο αυτό κάποιο που θα έχει τα προσόντα και την ικανότητα να διεκπαιρεώσει μια τόσο δύσκολη αποστολή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει η κυρία Σενίσιν για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά τον συνάδελφο Ρίτσαρτ Χόιτ για την ε, εξαιρετική και μεστή του έκθεση. Ε, δεν μπορούμε φυσικά να σχολιάσουμε όλα τα επιμέρους σημεία της έκθεσης, γι' αυτό θα επικεντρωθώ στα δικαιώματα των γυναικών που είναι σε ολόκληρη τον κόσμο τα πρωταρχικά θύματα της ε, διακριτικής μεταχείρισης, ε, υπόκειται εξευτελισμούς, ταπεινώσεις, βιοπραγίες. Νομίζω ότι η ισότητα των δύο φύλων και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων είναι σημαντικό ε, πρωτοβουλία και θα πρέπει να προάγουμε τέτοιου στόχου. Δεν μπορούμε να αντιμετωπίζουμε και να δεχόμαστε αντιμετώπιση των γυναικών ω πολιτών ε, δεύτερη κατηγορία. Ε, αυτό θα πρέπει να το λάβουμε υπόψη και στις διάφορε ενέργειές μα υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη δημοκρατία. Θα πρέπει να περιλάβουμε και την άσκηση βία κατά των γυναικών που μπορεί να είναι σωματική, ψυχολογική, κοινωνική, οικονομική και πολιτική. Θα πρέπει τα δικαιώματα των γυναικών να αποτελέσουν σημαντική προτεραιότητα στις διαπραγματεύσεις μας με τις υποψήφιες για ένταξη χώρες. Θα ήθελαμε να ε, επιθυμήσουμε στην Τουρκία ότι η καταπίεση των γυναικών, ακόμη και οι δολοφονίες λόγω τιμής, είναι σημαντικά εμπόδια του ενταξιακού δρόμου της ε, Τουρκίας. Επίσης, ε, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τις επιλεκτικές αμβλώσεις, ιδιαίτερα όταν το έβρινε και να προωθήσουμε πολιτικές ε, ε, για καλύτερη ενημέρωση ό,τι αφορά την αναπαραγωγική Αγία και την ισότητα των δύο φύλων. Αυτό θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα τη αναπτυξιακή πολιτική Ευρωπαϊκή Ένωση. Απευθύνουμε έκκληση προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τι ε, χώρε μέλη ώστε να πρωτοστατήσουμε στην πάταξη της βίας κατά των γυναικών ανά τον κόσμο και να συμπεριλάβουμε τη διάσταση της ισότητας των δύο φύλων στα ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει η κυρία Λουτφόρτ για μιση λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Χαίρομαι διότι στηρίζει ο εισηγητής την τροπολογία μου για την ανάγκη ευρωπαϊκής λογοδοσίας ε, για τα βασανιστήρια και τις ε, παραδόσεις, ούτως ώστε να παίξουμε ε, ένα θετικό ρόλο. Ελπίζω να γίνει δεκτή και ελπίζω όλοι να επικυρώσουν την σύμβαση για τις εξαφανίσεις. Για να απαντήσω σε μία η απάντηση σε μια γραπτή μου ερώτηση όμως δεν με ε, διαβεβαίωσε ότι ε, η ε, καταπολέμηση του λαθρεμπόριου ναρκωτικών στην Κεντρική Ασία είναι αποτελεσματική. Θα ήθελα να δοθεί συνέχεια στο ζήτημα αυτό. Πάντως είναι πολύ σημαντικό το θέμα των βασανιστήριων και το ρόλο των φαρμακευτικών προϊόντων και άλλων εργαλείων που εξάγονται και χρησιμοποιούνται κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταξύ άλλων και για τις ε, ε, ε εκτελέσεις. Θα ήθελα να πω στον Ρίτσαρντ Χάουιτ ότι ε, είναι πολιτική του Ηνωμένου Βασιλείου να ε, γίνει προσχώρηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ίσως ήταν κάπως αόριστη ε, σε σχέση με τις λεπτομέρειες. Αλλά από το Λονδίνο έμαθα ότι δεν υπάρχει καμία αντίρρηση ε, σε σχέση με μια ανάληψη δέσμευσης ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να προσχωρήσει στην σύμβαση αυτήν. Ευχαριστώ ο κύριος Στίβενσον για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Βαρώνει Άστον δεν θα εκπλαγείτε από το γεγονός ότι δεν μπορώ να αφήσω την ε, ευκαιρία να περάσει χωρίς να αναφέρω το στρατόπεδο Άσραφ ε, που ε, είχε προβλεφθεί ως προσωρινό κατάλημα για λίγες εβδομάδες Ορισμένοι έχουν μείνει τώρα τρεις μήνες εκεί και φαίνεται ότι θα αναγκαστούν να παραμείνουν στο στρατόπεδο αυτό για μήνες. Το στρατόπεδο αυτό, το καταβλισμός αυτός δεν επαρκεί για να καλύψει το μεγάλο αριθμό των προσφύγων που ζουν σε, ε, σε κατεστραμμένα κοντέινερ και δεν μπορούν ούτε να τα επισκευάσουν, ούτε μπορούν να ε, έρθουν ε, να έρθει βοήθεια, ε, ούτε μπορούν να γίνουν ε, υποτυπώδεις δρόμοι και μονοπάτια, ούτως ώστε άνθρωποι με ειδικέ ανάγκες να μετακινούνται. Και η κυβέρνηση του Ιράκ ε, πέτρεψε σε εκπροσώπους από το Υπουργείο Πληροφοριών στο Ιράν να εγκατασταθούν δίπλα στον καταβλισμό. Αυτό συνιστά παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Παρακαλώ, Βαρόνι Άστον, επιδείξτε πυγμή απέναντι στην κυβέρνηση του Ιράκ. Εξηγήστε τους ότι θα πρέπει να ε, ανταποκριθούν στα δίκαια αιτήματα των κατοίκων στο Άσραφ. Ευχαριστώ, ο κύριος Βανέκη, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Η έκθεση είναι ένα είδος καταλόγου καλών προθέσεων. Κάποιες ίσως είναι και λίγο αφελής, αλλά βασίζεται κατά κύριο λόγο στην ιδέα ότι αν ρίξουμε περισσότερα χρήματα σε διάφορες υπηρεσίες δημόσιες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα βελτιωθεί η κατάσταση σε ολόκληρο τον κόσμο. Ε, αυτό είναι λάθος. Ε, είναι αυτή η πολιτική ορθότητα που είναι το ε, ελάττωμα αυτής της έκθεσης. Ε, γίνεται μια αναφορά στα δικαιώματα των γυναικών και των ε, μειονοτήτων των θρησκευτικών στις Ισλαμικές χώρες. Αναφέρεται στο παράδοξο της Αραβικής Άνοιξης, όπως είναι γνωστή πλέον, αλλά πολύ προσεκτικά αποφεύγει να αναφέρει το Ισλάμ ως πρόβλημα. Και αυτό πιστεύω ότι είναι ο πυρήνας του προβλήματος. Ε, ζητάμε διάφορες ε, δράσεις ε, με σκοπό να διασωθούν οι λαθρομετανάστες με πολύ υψηλό τίμημα βεβαίως. Το δέχομαι αυτό, αλλά δεν αναφέρει τίποτα για την επαναπρόθεσή τους στις χώρες προελευσής τους, γιατί αυτό δεν είναι πολιτικά ορθό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Μπρόκ. Μπρόνς, με συγχωρείτε, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση για να είναι ένα αξιόπιτο παίκτη πρέπει να είναι συνεπή και να αποφεύγει ε, διαφορετικά μέτρα για σταθμά μεταξύ εσωτερική και εξωτερική πολιτική. Πρέπει η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση να εφαρμόζει ε, αυτά που καταδικάζει σε άλλου. Ε, οι τυραννίες ε, εμποδίζουν την ελευθερία έκφρασης αλλά ε, δεν θα πρέπει να ε, αναφερόμαστε στο τι γίνεται στην Τουρκία όταν η Γαλλία και άλλες χώρες πέρασαν παρόμοιες νομοθεσίες καθώς και άλλες χώρες. Η μη επιτυχής δίωξη του Γκίλ Βίντερς παραβλέφθηκε όταν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συζήτησε το θέμα της φυλάκη, τη θανάτια της του Βίλντερς για την ιστοσελίδα του. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να προσπαθήσει να ε, διαχύσει τα ανθρώπινα δικαιώματα έξω από τα σύνορά της, θα πρέπει να φροντίσει πρώτα τα του οίκου της. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Μπρόκ για 1,5 λεπτό. Κυρία Αντιπρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχήν ευχαριστήσω τον κύριο Χάουιτ για την εξαιρετική εργασία Θεωρητικά είμαστε σύμφωνοι σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το θέμα είναι πώς στην πράξη ε, θα τα υπερασπιστούμε και πώς θα λειτουργήσει η υπηρεσία εξωτερικής δράσης. Ενδεχομένως θα πρέπει να υπάρξει και ένα τμήμα που θα ασχολείται με τη θρησκευτική ελευθερία, γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό. Στην Αίγυπτο βλέπουμε τις εξελίξεις, βλέπουμε τους φόβους ε, των χριστιανών, ένα εκατομμύριο είναι έτοιμοι να φύγουν ή βλέπουμε την συνταγματική διαδικασία στην Αίγυπτο. Περίπου 15 εκατομμύρια κόπτες αντιμετωπίζουν τελείως διαφορετικά δεδομένα. Ε, γιατί υπήρξε ένα μόντους βιβέντι ε, με το ε, Ισλάμ. Τώρα όμως υπάρχουν ε, διαφοροποιήσεις που πρέπει να μας απασχολήσουν ιδιαίτερα για να προλάβουμε και κύματα μετανάστευσης. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα των διώξεων των χριστιανών. Επίσης πρέπει να εξετάσουμε τις εμπορικές συμφωνίες η συμφωνία, η συμφωνία σύνδεσης με την Ουκρανία ακόμη δεν έχει ε, υπογραφεί στο βαθμό που διώκονται μέλη της αντιπολίτευσης, στο βαθμό όπου ε, οι ασθενείς ε, βασική εκπρόσωπος της ε, ε, αντιπολίτευσης κρατείται ή στο βαθμό που χρησιμοποιούνται βασανιστήρια όπως διαπιστώνουν οι γιατροί. Θα πρέπει να πούμε ότι περιορίζονται όλες οι πρακτικές και στρατηγικές μας σκέψεις και δυνατότητες. Ε, όμως δεν θα πρέπει να κάνουμε πίσω στις θεμελιώδεις μας αρχές. Για 1,5 λεπτό κυρία Γκόμες. Ευχαριστώ. Ακούσαμε την ε, πολιτική δήλωση για τη νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τον ορισμό του ειδικού εντεταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Παρακαλώ λάβετε υπόψη τις ανησυχίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όπως εκφράζονται στην πολύ σημαντική έκθεση του Ρίτσαρτ Χάουιτ, του συναδέλφου τον οποίο και ευχαριστώ θερμά. Ε, Επίσης, θα ήθελα να ζητήσω από τους συναδέλφους της δεξιάς πτέρυγας να αναθεωρήσουν την ψηφοφορία, τη θέση τους στην ψηφοφορία ε, σε ό,τι αφορά την τροπολογία για την αναπαραγωγική υγεία και τα δικαιώματα των αποφυλοφίλων διεμφυλικών, ε, σε ό,τι αφορά επίσης τη, τους βασανισμούς ε, στις μυστικές φυλακές και τα εγκλήματα πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας θα πρέπει η προαγωγή της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να βρεθούν στο επίκεντρο της πολιτικής της ΕΕ. Θα έχουμε κάποια μαθήματα να διδαχθούμε από την Αραβική Άνοιξη και θα πρέπει να σταματήσει η στήριξη σε καταπιεστικά, κατασταλτικά καθεστώτα υπό το πρόσχημα της ασφάλειας, της σταθερότητας, των οικονομικών συμφερόντων Δείτε τι έγινε στην Αιθιοπία. το δικτατορικό αυτό καθεστώ είναι σημαντικό δικαιούχο τη αναπτυξιακή βοήθεια ε, τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, όταν έχουμε περισσότερα για περισσότερα να εφαρμόσουμε ταυτόχρονα και το λιγότερα για λιγότερα. Χρειαζόμαστε BFE και δραστήρια υποστήριξη τη κοινωνία των πολιτών, αν την υποστηρίζουμε κατασταλτικά και καταπιστικά καθεστώτα, να υποστηρίζουμε του φορεί του εκδημοκρατισμού. Ενώ ταυτόχρονα οι εμπορικέ και οικονομικέ μα πολιτικέ θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη και τι προσπάθειε σε δημοκρατία και ανθρώπινα δικαιώματα των εταίρων μα και το προσωπικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις αντιπροσωπείς μας, στα γραφεία μας και οι επικεφαλής αντιπροσωπείων μας θα πρέπει να έχουν ειδική εκπαίδευση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία. Η νέα στρατηγική θα πρέπει να τεθεί υπό κοινοβουλευτικό έλεγχο και τα διάφορα έγγραφα κείμενα θα πρέπει να διέρχονται από διαδικασία διαβουλεύσεων με την κοινωνία των πολιτών και να δημοσιεύονται. Ελπίζω, κυρία Άστον, όταν ε, επισκέφτεστε χώρες όπου οι ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων αντιμετωπίσουν προβλήματα, να έρχεστε σε επαφή μαζί τους και να λαμβάνετε υπόψη τον προβληματισμό και τις ανησυχίες τους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Κόβαλ για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε. Η πρώτη μου παρατήρηση ίσως είναι και πιο σημαντική. Πολύ συχνά μιλούμε για τις χώρες που διέρχονται από μεταρρυθμίσεις και σε μεταβατική διαδικασία. Μιλούμε για οικονομικές και άλλες μεταρρυθμίσεις. Είχαμε την φυλάξη της Τιμοσέγκο στην Ουκρανία. Πάντως πιστεύω ότι η βάση για την εξασφάλιση σωστής δημοκρατικής μεταρρύθμισης είναι η μεταρρύθμιση του δικαστικού κλάδου δεν μπορούμε να το παραμελούμε αυτό. Θα πρέπει η δικαστική μεταρρύθμιση να είναι ο γνώμονάς μας για την εξέταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ε, είμαι υπέρ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Δημοκρατίας, αλλά φοβούμε μήπως ακόμη και στα σπάργανά του πνιγεί στην γραφειοκρατία αυτό το ταμείο. Θα πρέπει να υποστηρίξουμε τη δημοκρατική διαδικασία στη Λευκορωσία, στην Βόρεια Αφρική, αλλά να περιορίσουμε τη γραφειοκρατία για να δώσουμε ε, μεγαλύτερη όθηση στο ταμείο αυτό μια πολύ σημαντική έκκληση. Ας μην φοβηθούμε να πούμε ότι η πιο διοκόμενη και καταπιεσμένη ομάδα είναι η, μειονότητα, η χριστιανική μειονότητα σε πολλές χώρες. Νομίζω ότι για να ε, γίνουμε αξιόπιστοι θα πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, να λέμε τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη και να μην φοβόμαστε να κάνουμε τέτοιες δηλώσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Προβέρα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρία Άστον. Η ελευθερία της θρησκείας φαίνεται να κινδυνεύει όλο και περισσότερο και ιδιαίτερα διαδίονται όλο και περισσότερο περιπτώσεις δίωξης ε, των χριστιανών στη Μέση Ανατολή, στην ε, Αφρική κατά του ιδιαίτερα στην Ιγυρία, στην Νοτιοανατολική Ασία, στην Κίνα, στην Ινδία, στο Πακιστάν και στην Βόρεια Κορέα. Στι χώρε αυτέ είναι πάρα πολλέ οι περιπτώσει τη εξαναγκασμένη μετανάστευση, ε, των επιθέσεων, ε, των βασανιστήριων, των δολοφονιών και εξαναγκαστικών προσλητισμών. Τουλάχιστον 10% των χριστιανών σε ολόκληρο τον κόσμο Δηλαδή 200 εκατομμύρια άνθρωποι είναι μειονότητες στις χώρες τους και δυνάμει θύματα διακριτικής μεταχείρισης. Η θρησκευτική ελευθερία είναι ένα θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα, όλοι το γνωρίζουμε αυτό, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι διεθνείς οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα δυστυχώς είναι ακόμα πολύ λίγο αποτελεσματικές στην ε, ε καταγγελία και στην προστασία του δικαιώματος αυτού. Και με την ευκαιρία αυτή προτείνω και πάλι ε, να υπάρχει μια ε, επικαιροποιημένη αιτήσια έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα παρακολουθεί την κατάσταση της θρησκευτική ελευθερίας σε ολόκληρο τον κόσμο και όπου θα καταδικάζει έντονα τις παραβιάσεις του όπου υπάρχουν αυτές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει... Ε... Για 1,5 λεπτό ο κύριος Βαγουένσα. Ευχαριστώ. Κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Χάουιτ για την έκθεσή του που είναι πολύ καλό σημείο αφετηρία ε, για το δύσκολο αυτό θέμα. Ε, με εξαντλητικό τρόπο μιλάει για το θέμα αυτό στα πλαίσια της πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης η έκθεση Χάουιτ. Ε, γίνονται ε, κάποιες παρατηρήσεις ε, για την οικονομική κρίση και για την ανεργία και είναι εύκολο μερικές φορές να ξεχνούμε σημαντικές αξίες όπως είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα. Βέβαια, η υλοποίηση αυτών των αρχών και αξιών θα πρέπει να αποτελέσει σίγουρα θεμελιώδη ε, θεμελιώδη προϋπόθεση που θα πρέπει να τηρούν χώρες που προσβλέπουν σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό θέμα και δεν μπορούμε να το ε, παραβλέπουμε. Ούτε θα πρέπει να ε, θυσιάζουμε στο βωμό οικονομικών δικαιωμάτων κάποια δικαιώματα ατόμων ή ε, μειονοτήτων ή κοινοτήτων. Ο προβληματισμός αυτός είναι πολύ επίκαιρος γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε εμπορικές αλλά και ενταξιακές διαπραγματεύσεις με χώρες που δεν ευθυγραμμίζονται σε ό,τι αφορά τη δική μας ερμηνεία και αντίληψη για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά τα παραβιάζουν συστηματικά. Ε, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να μετατραπεί σε παγκόσμιο θεματοφύλακα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Έχουμε όμως αρκετούς αποτελεσματικούς μηχανισμούς, ιδιαίτερα στη συνεργασία μας με τις τρίτες χώρες για να προσπίσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Νομίζω ότι αυτό θα πρέπει να είναι η υψηλή μας προτεραιότητα σε όλες τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κάνω ένα βήμα προς τα πίσω. Κύριε Προβέρα, δέχεστε μία ερώτηση με μπλε κάρτα από τον κύριο Δεκέιζερ. Παρακαλώ. Είναι Ευχαριστώ. Δεν είναι αρνητική ούτε ε, κακή η κάρτα μου. Όταν μιλάτε για αναξιθρησκεία και θρησκευτική ελευθερία, εγώ είμαι αγνωστική ίστρια. Γιατί να μιλούμε και για την ε, ελευθερία πεπιθήσεων ε, γιατί όταν ζητάτε έκθεση για την ανεξιθρησκεία ή για το δικαίωμα θρησκευτικής ε, λατρείας ή θρησκευτική ελευθερία, έχω την αίσθηση ότι ακροτηριάζουμε την συνέλευση από τους μισούς ίσως ή συμμετέχοντες από τα μισά μέλη. Ναι, κύριε Προβέρα. Είμαι υπέρ αυτής της έκθεσης, αλλά αφήστε και σε εμά τους α, ε, α, ε, μη πιστεύοντες, τους λαϊκούς, να εκφράσουμε τη φιλοσοφία μας για τη ζωή, την κοσμοθεωρία μας, ε, τον τρόπο που αντιμετωπίζουμε την πνευματικότητα, που μπορεί να μην ευθυγραμμίζεται με το δικό σας, γιατί με τέτοια μονομερή σχόλια αισθάνομαι προσβεβλημένη και Ιδιαίτερα με ενόχλησε η δρυμύτατη επίθεση κατά του Ισλάμ από ένα συναδελφό σας. Παρακαλώ. Αυτό που επιθυμώ εγώ να γίνει είναι μια λεπτομερής έκθεση για οποιαδήποτε παραβίαση της ελευθερίας της λατρείας, όπου για να συμβαίνει αυτή και για όποια θρησκεία και να πρόκειται. Ε, όποια θρησκεία και να είναι αυτή που απαγορεύεται να ασκείται σε οποιοδήποτε σημείο του κόσμου. Δεν υπάρχει καμία διάκριση εις βάρος οποιασδήποτε θρησκείας. Είναι μια έκθεση που ε, βασίζεται σε κάποιες διαπιστώσεις, δηλαδή από τις 300 ε, ε, επιθέσεις που γίνονται εναντίον των χριστιανών σε ολόκληρο τον κόσμο που είναι όλο και πιο σοβαρές και όλο και πιο συχνές. Εγώ λοιπόν θεωρώ ότι εφόσον αυτό εδώ το κοινοβούλιο θεωρεί ότι είναι θεμελιώδης η προστασία όλων των δικαιωμάτων του ανθρώπου, ίσως το θρησκευτικό δικαίωμα είναι το πιο θεμελιώδες γιατί ξεκινάει από από μια ηθική απέτηση και όχι μόνο από μια ανθρώπινη ανάγκη. Και θα πρέπει να το υπερασπιστούμε το δικαίωμα αυτό, γιατί έτσι είμαστε συνεπείς και προς τις αρχές αυτού του Κοινοβουλίου και προς την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που πολλές φορές χαιρετίζονται ως ε, μια ε, κατάκτηση της ανθρωπότητας. Ε, e Ευχαριστώ για ένα μισή λεπτό. Η κυρία Ντεκέιτσερ. έχει το λόγο. Θα πάω να πιω ένα καφέ με τον κύριο Προβέρα για να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση. Αλλά πιο σοβαρά. Ε, δύο λόγια για την έκθεση του Ρίτσαρντ Χάουιτ που θεωρώ ότι είναι εξαιρετική και που δεν χρειάζεται καθόλου τρόπο πιστεύω. Αλλά ήθελα να αναφερθώ σε δύο σημεία. Το ένα είναι η υπεράσπιση των γκέι και των λεσβιών που κρύβεται, έχει αποκριθεί κάπου μέσα στη νέα διατύπωση και αυτό είναι λυπηρό. Η κυρία Άστον και η ε, Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης όλοι θα πρέπει να φροντίζουμε ώστε στις εταιρικέ μας σχέσεις να γίνονται απολύτως σεβαστά τα δικαιώματα των ε, ομοφιλόφιλων και των λεσβιών. Είναι τεράστια δουλειά που πρέπει να γίνει στο επίπεδο και σας παροτρύνω κυρία Άστον να αναλάβετε δράση. Το δεύτερο σημείο στο οποίο θα ήθελα να επανέλθω είναι η περίφημη νέα πολιτική γειτονία και το περισσότερα για περισσότερα. Έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στο Συμβούλιο, στην Οικομισιόν, στις υπηρεσίες σας. Έχουμε όμως παρόλα αυτά τον φόβο ότι αυτή η νέα πολιτική γειτονίας θα ε, παραμείνει εξίσου τυφλή μερικές φορές απέναντι στην πραγματικότητα των χωρών όταν ε, έχουμε σχέσεις ε, με αυτές τις χώρες όταν είναι συμμαχοί μας όπως ήταν και η παλιά. Και αυτό θέλουμε να κάνουμε πιο λειτουργικό. Ο Ρίτσαρντ, είπε πολύ σωστά ότι θέλουμε μια μέθοδο, θέλουμε κριτήρια, θέλουμε να μπορούμε να μετρήσουμε τις βελτιώσεις όσον αφορά τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα πραγματικά περισσότερα για περισσότερα. Αλλά ποιο μπορεί να το μετρήσει αυτό, ποιο μπορεί να το ζυγίσει. Αυτό είναι το πραγματικό ζήτημα. Και εδώ ε, υπάρχει μια πραγματική βούληση για αλλαγή που θα διαβεβαιώσει, θα επιβεβαιώσει το Κοινοβούλιο με την ψήφο του για την έκθεση αυτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κύριος Πόσελτ για 1,5 λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, η Λέδη Άστον έχει δίκιο από τις πρώτες άμεσες εκλογές του 1979 το Ευρωκοινοβούλιο συστηματικά ασχολείται με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το ίδιο θέλουμε να κάνουν το Συμβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και εδώ είστε εσείς υπεύθυνοι. Η Εδώ βρίσκεται και η σημασία της σημαντικής ε, συζήτησης. Ε, διώξεις χριστιανών. Κυρία Ντεκάιζερ, έχετε δίκιο. Η θρησκευτική ελευθερία ε, ε, πρέπει να περιλαμβάνει αγνωστικιστές. Όμως οι χριστιανοί σε όλο τον κόσμο διώκονται με έναν εντελώς ιδιαίτερο ε, τρόπο και η Ευρώπη, η χριστιανική κυρίως Ήπειρος, θα πρέπει να το λάβει αυτό υπόψη της. Θα πρέπει να είναι ο υπέρμαχος και ο προστάτης των χριστιανών σε όλο τον κόσμο. Το, ε, βεβαίως θα πρέπει να προστατεύονται οι ομοφιλόφιλοι, ε, αλλά θα αναφέρομαι και τους χριστιανούς. Είναι ιδιαίτερη ομάδα στόχος στην πολιτική ανθρωπίνων δικαιωμάτων οι χριστιανοί. Επίσης χρειάζονται τα ίδια μέτρα και σταθμά για όλους. Δεν μπορεί να επικρίνουμε τις ε, μικρές χώρες και να εξαιρούμε την Κίνα ή τη Ρωσία. Τα αυστηρά κριτήρια θα πρέπει να είναι τα ίδια για τους μεγάλους όπως και για τους μικρούς παρόλα τα οικονομικά συμφέροντα που ίσως θίγονται. Τρίτον και τελευταίο, είναι σημαντικό τα ανθρώπινα δικαιώματα να μην ε, αντιμετωπίζονται καταχρηστικά. Θα πρέπει να ισχύουν για όλους τους ανθρώπους. Η κατάχρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, για να επιβληθούν συγκεκριμένες απόψεις ε, δεν ε, ε, ταιριάζει και στο, στο, ήθος και στη μέχρι τούδε πρακτική του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Κύριε Πόσελτ, δέχεστε μια γαλάζια κάρτα από τον κύριο Βάιγκλ. Βεβαίως, λέει ο κύριος Πόσελτ. Είμαι πεπισμένος ότι ο κύριος Πόσελτ θα απαντήσει δημιουργικά στην, ερώτησή μου. Δεν πιστεύει ότι στην Ευρώπη θα γίνουμε πιο αξιόπιστοι αν βοηθήσουμε τους χριστιανούς σε όλο τον κόσμο και αν με την ίδια προσοχή παρακολουθούμε και τα δικαιώματα και την ε, αξιοπρέπεια άλλων θρησκευτικών μειονοτήτων που ζουν στο δυτικό ημισφαίριο και την Ευρώπη. Πολλές φορές ε, εκπρόσωποι άλλων θρησκείων ε, ενοχλήθηκαν και δικαίως λόγω των καταχρηστικών πρακτικών σε βάρος των θρησκευτικών τους ε, αισθημάτων. Κυρία Πρόεδρε, μιλάμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο, εκτός Ένωσης και υπάρχει ένα ιδιαίτερο πρόβλημα των διώξεων των χριστιανών. Φυσικά και θα πρέπει να βοηθήσουμε και να υπερασπιστούμε μουσουλμάνους σε όλο τον κόσμο. Οι διώκονται στη Σερβία, για παράδειγμα, οι μουσουλμάνοι που είναι και υποψήφια χώρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι τεράστιο το πρόβλημα σε κάποιες περιοχές εκεί και σε πολλές άλλες. Και βέβαια είναι απαραβιέστια η ανθρώπινη αξιοπρέπεια ανεξάρτητα από την γνώμη που θα εκφράσει ή τη θρησκεία ε, που πιστεύει. Ευχαριστώ, ο κύριος Κοστέλο, για ένα λεπτό. Η κυρία. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καλωσορίζω την έκθεση αυτή και θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή τον κύριο Ρίτσαρτ Χάουιτ. Υπάρχουν δύο θέματα στα οποία θα ήθελα να αναφερθώ από την έκθεση αυτή. Πρώτα απ' όλα το θέμα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να επιδιώξει την λογοδοσία για παραβίαση του διεθνού δικαίου. Και επ' αυτού θα ήθελα να υποστηρίξω πλήρω την τροπολογία που υπάρχει σχετικά με την Γάζα και τα κατεχόμενα. Όπως Υπόθηκε προηγουμένω και το έχω πει και εγώ. Ε, πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δείξει συνέπεια ανάμεσα στι πολιτικέ μα και τα ψηφίσματά μα αφενό και τι εξωτερικέ μα σχέσει και τη διμερεί συμφωνίε εφετέρου. Δεύτερον, τα θέματα, το θέμα των δικαιωμάτων ε, των ομοφυλόφιλων, λεσβιών κλπ. και τη ταυτότητα του φύλου. Θα ήθελα να υποστηρίξω τι τροπολογίε 7 και 8 που ενισχύουν την ε, έκθεση ε, από την άποψη αυτή. Θα πρέπει να φύγει η ταυτότητα του φύλου από την κατηγορία των διαταραχών, των διανοητικών διαταραχών. Πολλές φορές αυτό εμποδίζει ε, την ε, ε, έκδοση διαβατηρίου σε σχέση με την ταυτότητα του φίλου και αυτό είναι φυσικά μια κατάφορη παραβίαση των δικαιωμάτων των ανθρώπων αυτών. Το λόγο έχει για 1,5 λεπτό ο κύριος Μιγιάν Μον. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχήν κυρία Άστον, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω για τα σχόλια σας ό,τι αφορά την παράνομη και αυθαίρετη εθνικοποίηση της Ρεψόλ. Είναι ένα μέτρο που επηρεάζει όλους τους Ευρωπαίους και κατάφορα παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Σας ευχαριστώ και πάλι για τα σχόλιά σας. Ό,τι αφορά την έκθεση Howitt, τα άρθρα 3 και 21 της για την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, αναδεικνύουν την τεράστια σημασία των, ευρωπαϊκών δικαιωμάτων, των ε, ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μάλιστα το κράτο δικαίου και τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν ακρογωνίου λήθου ε, των κρατών μελών και τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και μάλιστα τη σήμερα ημέρα η σύσσωμη διεθνή κοινότητα θεωρεί ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι αδιέρετα, αναπαλωτριώτα και οικουμενικά. Και σίγουρα δεν θα πρέπει από το πρόσχημα της μη επέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις μιας χώρας ε, να μην ε, υποστηρίζουμε και να μην υπερασπίζουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι σημαντική η θέση που έχουν τα ανθρώπινα δικαιώματα για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ενδεικτικό είναι το βραβείο Ζαχάροφ που θεσπίσαμε υπέρ αυτών και νομίζω ότι είναι ε, συμβολική και η πρόταση για, το διορισμό ειδικού εντεταλμένου τη ευρωπαϊκή Ένωση ενό είπα το ορμοστή για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το θέμα είναι πολύ επίκαιρο. Έχουμε ε, σίγουρα ένα καινοτόμο θεσμό επιφορτισμένο με την ε, ανάγκη πρόσβησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και είχαμε και τα πρόσφατα γεγονότα της Αραβικής Άνοιξης που είχε προδοχικό στόχο την διάσωση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα πρέπει οι νέες πολιτικές μεταρρυθμίσεις ε, να εμπεδώσουν ε, τις ε, απαιτήσει για δημοκρατία, ανθρώπινα δικαιώματα και να μην τι διακυβεύσουν, γιατί και το δικαίωμα των μειονοτήτων είναι ένα από τα σημαντικά ανθρώπινα δικαιώματα. Το λόγο έχει η κυρία Παπαδοπούλου για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Στον απόϊχο της Αραβικής Άνοιξης η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να διδαχθεί από λάθη του παρελθόντος. Να μην εφαρμόζει πολιτικές δύο μέτρων και δύο σταθμών. Σωστά προτάσει στον πυρήνα της εξωτερικής της πολιτικής, τον έλεγχο της εφαρμογής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τον εκδημοκρατισμό στι δράσεις τρίτων χωρών. Ωστόσο, δεν πρέπει να εθελοτυφλεί όταν εντό τη ίδια τη Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν χώρε όπου η Κύπρο, όπου τα ίδια ανθρώπινα δικαιώματα παραβιάζονται από την κατοχική τουρκία χωρί τιμωρία. η ευρωπαϊκή ένωση οφείλει να επιβάλλει ρήτρε προστασία και εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε όλε τι εμπορικέ και τομεακέ συμφωνίε με τρίτε χώρε, να επιβάλλει κυρώσει καταργώντα διακρίσει κατά γυναικών και μειονοτήτων να τερματίσει διώξει εναντίον βουλευτών συνδικαλιστών και δημοσιογράφων στην τουρκία να καταπολεμήσει την ατιμορρησία αξιοποιώντα το διεθνέ ποινικό δικαστήριο να οικοδομήσει μέσω τη παιδεία μια πραγματική κουλτούρα σεβασμού στα ανθρώπινα δικαιώματα. τέλο οφείλει να ενισχύσει το ρόλο του ευρωκοινοβουλίου τη λογοδοσία και διαφάνεια και να εξεύρει αποτελεσματικού μηχανισμού εφαρμογή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παντού. Ευχαριστώ. Δέκα ε, συνάδελφοι έχουν ζητήσει να μιλήσουν στη διαδικασία Catch Θα δώσω το λόγο σε όλους, αν, διατηρήσετε, αν τηρήσετε όμως το χρόνο του ενός λεπτού. Μια στιγμή παρακαλώ. Κυρία Παπαδοπούλου, δέχεστε μια ερώτηση βλεκάρτας. Ο κύριος Πόσελτ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ρωτήσω την κυρία Παπαδοπούλου αν θα φροντίσει και εκείνη ώστε η Κυπριακή Προεδρία που την περιμένουμε με χαρά με σαφέστερο τρόπο θα υποδείξει στην Τουρκία το θέμα της στήριξης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μίλησε καθαρή γλώσσα και κυρία Άστον χρειάζεται η ίδια σαφής γλώσσα από το Συμβούλιο και την Κομισιόν. Και θα μπορούσε εδώ η συνάδελφος κυρία Παπαδοπούλου να μας βοηθήσει σε σχέση με την Κύπρο.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 η θέση της κυπριακής δημοκρατίας είναι απόλυτα ξεκάθαρη. η κύπρος δεν έχει ασκήσει κανένα βέτο για την ενταξιακή πορεία της τουρκίας. η τουρκία ωστόσο οφείλει να υλοποιήσει το πρωτόκολλο της άγκυρας να αναγνωρίσει την κυπριακή δημοκρατία και να σταματήσει τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην κύπρο. εάν πράξει όλα αυτά που είναι υποχρεώσεις μιας χώρας υποψήφιας προς ένταξη απέναντι στην ευρωπαϊκή ένωση η κύπρος δεν έχει κανένα πρόβλημα να κάνει ό,τι πρέπει όσον αφορά την ενταξιακή πορεία της Τουρκίας. Επομένως, η μπάλα είναι στο γήπεδο της Τουρκίας. Ευχαριστώ. Catch the eye. Γκάλ. Κυρία Γκάλ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Ήπατη εκπρόσωπε, πέρσι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ασχολήθηκε με την ετήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα που αποτέλεσε ένα σημαντικό μέσον. Όλοι την παρακολουθούν εντός και εκτός Ευρώπης και οι τρίτες χώρες ενδιαφέρονται για την έκθεση αυτή και το περιεχόμενό της είναι πολύ σημαντικό. Η ποιότητα επίσης. Συγχαίρω τον κύριο Χάουιτ για την εξαιρετική του έκθεση. Μια έκθεση που είναι αξιοπρόσεκτη σε σχέση με αυτά που είπε η υπατή εκπρόσωπος. Ωραία είναι τα λόγια, ακόμα καλύτερα τα έργα. Θα πρέπει να ενισχύσουμε την βοήθεια της διατιθέμενης βοήθειας. Τα μέσα προώθησης αναφέρθηκαν, τα ταμεία, τα ταμεία όμως θα πρέπει να έχουν συγκεκριμένη επίπτωση θετική στα ανθρώπινα δικαιώματα όταν αυτά καταπατούνται. Ε, θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας στο γεγονός ότι υπάρχουν κοινότητες, εθνοτικές μειονότητες, παιδιά ε, που είναι ευάλωτοι. Ακούσαμε για όλες τις κοινότητες αυτές. Αυτοί είναι που ε, υποφέρουν πιο πολύ. Ματέρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, η έκθεση αποτελεί μια ετήσια αξιολόγηση του πόσο οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης είναι προσανατολισμένες προς τα ανθρώπινα δικαιώματα σε ολόκληρο τον κόσμο. Είμαι υπέρ μιας κριτικής προσέγγισης, αλλά ταυτόχρονα επικοδομητικής όσον αφορά την ενίσχυση των πολιτικών υπέρ της ε, προώθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των γυναικών που πολύ συχνά αποτελούν μια αδύναμη ε, ε μειονότητα χωρίς ε, ε, ε χέγγια. Σε πολλές χώρες του κόσμου οι γυναίκες είναι η κύρια πηγή εισοδήματος για τις οικογένειες και για την οικονομία. Υπάρχουν διεθνείς οργανώσεις που ασχολούνται με αυτόν τον προβληματισμό και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να συνεργαστεί μαζί τους και μέσω ε, στοχευμένης χρηματοδότησης όπως μέσω του Trust Fund των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών. Καμία μορφή ε, των γυναικών δεν μπορεί να δικαιολογηθεί ε, στη βάση παραδόσεων, πολιτιστικών ε, κλπ. Και θα ήθελα να παρακαλέσω την κυρία Άστον ε, να κάνει κάτι για τους δύο ε, Ιταλούς ε, πεζοναύτες για το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Ο κύριο Σιλβέστρε. Ευχαριστώ. Ε, όλοι συμφωνούμε ότι είναι καλή αυτή η έκθεση. Δεν θα μπορούσε να είναι και διαφορετικά. Όλοι με τη σειρά μα υπογραμμίσαμε ε, ότι υπάρχουν δικαιώματα που παραβιάζονται, υπάρχει βία και διακρίσει ει βάρος των γυναικών, των ομοφυλόφιλων ε, με βάση θρησκευτική κλπ. Εγώ θα ήθελα να δώσω έμφαση, κυρία Άστον, σε μια κατηγορία που από την Ευρώπη δεν τη χάνει καμιά προσοχής. Εγώ εγώ υπέβαλα γραπτή δήλωση μαζί με άλλους συναδέλφους για να ε, δώσω ε, την ε, έμφαση στο πρόβλημα των ε, αμβλώσεων, των παιδιών που ποτέ δεν βλέπουν την ζωή για διάφορα προβλήματα που έχουν οι μητέρες τους. Το δικαίωμα στη γέννηση ε, είναι ένα θέμα το οποίο λείπει από τη συζήτηση αυτή. Ήθελα να ρωτήσω, σε πόσα χρόνια, σε πόσες δεκαετίες, σε πόσους αιώνες στην Ευρώπη θα εξεταστεί ε, το ενδεχόμενο και μόνο ε, να συζητηθεί το δικαίωμα της γέννησης πράγμα το οποίο σε άλλα σημεία του κόσμου γίνεται σεβαστό και εδώ το αρνούμαστε τόσο συχνά στην Ευρώπη. Κούγκαν. Ευχαριστώ. Συγχαρητήρια στον Ρίτσαρντ Χαούιτ για την σκληρή δουλειά και την εξαιρετική συνεργασία με συναδέλφους όδης που κατέληξαν στην ωραία έκθεση που έχουμε μπροστά μας. Τα ανθρώπινα δικαιώματα ήταν το ε, ήταν εδώ και καιρό το επίκεντρο της συζήτησής μας. Υπάρχει η γενική συμφωνία ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα και η δημοκρατία θα πρέπει να βρίσκονται στην καρδιά των εξωτερικών και εσωτερικών πολιτικών της Ένωσης. Πρέπει λοιπόν η ετήσια έκθεση να αφιερώνει σημαντικό κομμάτι για να ε, ενισχύει τη σύνδεση μεταξύ των δύο από το παρελθόν είδαμε ότι μόνο όταν έχουμε συνεπείς πολιτικές για τον εκδημοκρατισμό και την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μπορούμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνουμε διαφορά στις εξωτερικές δράσεις. Χαίρομαι διότι έχει μια εντρεωμένα θέση η, η Ευρωπαϊκή Ένωση ως προς την θανατική ποινή και καλό την είπα τη εκπρόσωπο να χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα πολιτικά μέσα για να ασκήσει πίεση στις χώρες που έχουν τη θανατική ποινή να την καταργήσουν ή να εφαρμόσουν εφαρμόσουν δικαιοστάσιο στην ε, εκτέλεση της ποινής αυτής, όπως η Λευκορωσία. Ο κύριος Μπαζέ. Κύριε Μπασέσκου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, θα ήθελα να πω ότι προκειμένου να προαγάγουμε αποτελεσματικά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία ανά τον κόσμο, χρειαζόμαστε αυτά μέτρα και δράσει. Γι' αυτό και συμφωνώ με το άρθρο 8 για τη θέσπιση σαφών κριτηρίων προκειμένου να αποτιμήσουμε την πρόοδο στο τομέα αυτό. Ας μην ξεχνούμε και την κατάσταση των κατοίκων στις περιοχές των παγωμένων συγκρούσεων τα δικαιώματα αυτών των ανθρώπων θα πρέπει να τύχουν κάποιες προστασίες και θα ήθελα να ζητήσω από την ΕΠΑΤΗ εκπρόσωπο επιπλέον προσπάθειες και επίτεση των ενεργειών για να εξασφαλιστούν αυτά τα δικαιώματα. Έχουμε και την ε, υπερδνηστερία. Πριν από λίγες μέρες είχαμε νέα επεισόδια στο Βάντε ε, στο φυλάκιο αυτό ελέγχου δεν θα πρέπει να ανεχόμαστε κατάφορη παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απαιτώ λοιπόν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο να, ε, ε, λάβουν, να αναλάβουν μέτρα προκειμένου να τιμωρηθούν ε, όσοι υποβάλλουν μισαλόδοξα και ξενοφοβικά σχόλια μέσω της Ολλανδικής ιστοσελίδας στις κατοχώρες. Η κυρία Τσικάου, ευχαριστώ. Το Ευρωπαϊκό Μέσο για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα αντανακλά τη δέσμευση τη Ευρωπαϊκή Ένωση για προώθηση και προαγωγή τη δημοκρατία και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στηρίζοντα ταυτόχρονα την κοινωνία των πολιτών, αλλά και φορεί και θεσμού που προσπίζουν τον κόσμο τα ανθρώπινα δικαιώματα. Για την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε χρηματοδότηση 1,4 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ είχαμε αρχικά 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Θα ήθελα να μιλήσω και για την τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών. Πολύ σημαντική η χρήση της για την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα πρέπει να προασπίσουμε και την ελευθεροτυπία και την ελευθερία έκφρασης, να υπερασπίσουμε τους δημοσιογράφους και τους bloggers, να εξασφαλίσουμε ελεύθερη πρόσβαση στην πληροφορία και την επικοινωνία και χωρίς λογοκρισία πρόσβαση στο διαδίκτυο. Επίσης θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και την ισότητα των φύλων και να εμπλέξουμε και τις γυναίκες στη διαδικασία επίλυσης των διαφορών. Ευχαριστώ. Η κυρία Μπένοβα. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, Άστον, αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να συγχαρώ τον Ρίτσαρντ Χάουιτ για την εξαιρετική έκθεση που κατέθεσε και αναδεικνύω το γεγονός ότι όταν μιλάμε για ανθρώπινα δικαιώματα παγκοσμίω, όταν αναφερόμεθα επίσης στις πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ, πέρα από τα θέματα που αναφέραμε, πρέπει να προσθέσουμε και τα κοινωνικά δικαιώματα. Τα κοινωνικά δικαιώματα θεωρούνται θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών μας και καταβάλω κάθε προσπάθεια, θα καταβάλω κάθε προσπάθεια για να τα ενσωματώσω στην έκθεση ως ανθρώπινα δικαιώματα. Σήμερα, εμεσούσεις της κρίσης και της ανεργίας, όταν μιλούμε για νόμιμους και παράνομους μετανάστες που εισέρχονται στο έδαφος της Ένωσης λόγω κοινωνικών προβλημάτων, πιστεύω ότι αυτή είναι μια κατάσταση που απαιτεί να δοθεί μεγαλύτερη σημασία στα κοινωνικά δικαιώματα που πρέπει να αντικατοπτρίζονται σε όλες τις πολιτικές της Ένωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Βάγκλ. Ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Εξαιρετική βέβαια η έκθεση του κυρίου Χάουιτ, αλλά δεν μπορεί να καλύψει όλες τις περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Νομίζω όμως ότι είναι σωστό να αναφέρομαι μια συγκεκριμένη παραβίαση που υπάρχει εδώ και δεκαετίες στη Δυτική Σαχάρα. Ο τρόπος ζωής σε καταβλισμούς προσφύγων είναι απαράδεκτος. Πρέπει λοιπόν να το αναφέρουμε το πρόβλημα αυτό και παράλληλα να προτείνουμε μια λύση που θα μπορέσει να εφαρμοστεί. Κυρία Άστον, θα ήθελα να σας πω ότι 83 πολιτικοί ε, κρατούμενοι από τη Δυτική Σαχάρα είναι σε μαροκινό έδαφος και στο Συμβούλιο Ασφαλείας ε, γίνεται συζήτηση για την αποστολή Μινούτσιο που είναι η μοναδική αποστολή που δεν έχει ε, δικαίωμα να παρακολουθεί τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και αυτό θα πρέπει να αλλάξει. Είχαμε μιλήσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, λέει κυρία Γιατερμάκη, για την ε, Κίνα και την κατάσταση των Ουιγούρων ε, στην πόλη Κασκαράρη. Και μάλιστα στη συζήτηση εκείνη, ο εκπρόσωπο τότε τη ε, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική Δράση διαπίστωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε ό,τι μπορούσε για να προασπίσει τα δικαιώματα αυτής της κοινότητας ε, και αυτή την περιοχή. Θα πρέπει λοιπόν να τηρήσουμε τις υποσχέσεις που δώσαμε ε, και να δώσουμε μια συνέχεια στο έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και να ενημερωνόμαστε τακτικά. Τι κάνατε κυρία είπατε εκπρόσωπε ώστε η πόλη Κασκαράη να αναδειχθεί σε παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO και να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα το, της κοινότητας των Ουιγούρων. Γίνονται όντως κάποιες προσπάθειες να υπερασπίσουμε αυτή την κοινότητα ή ήταν απλώς ε, επεπτερόεται υποσχέσεις σας. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει η ηταν απλως τα Λόχμπίλερ. Κυρία Πρόεδρε, κυρία Ήπατη εκπρόσωπε, αγαπητοί συνάδελφοι, η έκθεση αυτή για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ένα καλό κείμενο και ελπίζω ότι αυτή τη βδομάδα θα το εγκρίνουμε. Αναφέρομαι στις διαφορές απόψεων που είχαμε και έχουμε στο Κοινοβούλιο σε σχέση με αιτήματα που αφορούν διαφωτισμό, σε διαφώτιση σε σχέση με ανθρώπινα δικαιώματα όπως δημιουργία μυστικών φυλακών ή μυστικές παραδόσεις. Αυτό ε, ε, είναι πρόβλημα στην Ευρώπη. Πρέπει λοιπόν να το παρακολουθήσουμε, αλλιώς θα είμαστε αναξιόπιστοι ε, στην Ευρώπη. Πρέπει να αναφερθούμε στις υποχρεώσεις συγκεκριμένων κρατών μελών. Την περασμένη εβδομάδα διοργανώθηκε μια εκτενής ακρόαση πάνω στο θέμα αυτό. Παρακαλώ τους αναποφάσεις τους συναδέλφους να ψηφίσουν υπέρ των αιτημάτων αυτών, να έχουμε το θάρρος δηλαδή να αναπτύξουμε μια πολιτική η οποία θα αποτρέπει από τέτοια εγκλήματα στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία ε, ε, Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ και εσάς Λεδη Άστον για τα σχόλια που εκάνατε ήδη για την έκθεση. Ευχαριστώ και τον συνάδελφο Χάουιτ για την πολύ καλή έκθεση. Ένα θέμα θα ήθελα να αναφέρω και έγινε δεκτό από την Επιτροπή Αστροπολογία, δηλαδή ε, μηχανισμοί διαβούλευση τη κοινωνία των πολιτών που θα δημιουργηθούν σε σχέση με όλα τα μέσα που διαθέτουμε. Συγκεκριμένα αναφέρομαι στι δύο τροπολογίε που κάποιοι από εμά θα καταθέσουμε πάλι για την αυριανή ψηφοφορία. Είναι οι τροπολογίε 7 και 8 για του ε, λεσβείε, ομοφυλόφιλου, αμφίφιλους, ε, τρανσεξουαλικού. Ω λεσβεία έχω δει πολλά πράγματα στον κόσμο. Έχω δει περιπτώσεις ανθρώπων που δεν μπορούν ε, να, λειτουργήσουν ελεύθερα στις κοινωνίες τους. Καλό όλους τους ε, συναδέλφους που κατεψήφισαν ε, το σχετικό εδάφιο να ψηφίσουν υπέρ των τροπολογιών γιατί είναι, αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα τα κοινά, αφορά τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που όλοι προσυπογράφεται και που αναφέρει ότι δεν πρέπει να υπάρχουν διακρίσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρακαλώ ψηφίστε τις τροπολογίες, στηρίξτε ε, τα μέσα που διαθέτει η Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και η Λέδη Άστον, ούτως ώστε οι λεσβείες, οι αμφιφυλά, άτομα, ομοφυλόφιλοι και τρανσεξουαλικοί να ζουν χωρίς φόβο σε αυτή την κοινωνία. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μιράντα. Ευχαριστώ. Ήταν ε, πολύ άμεση και κατηγορηματική η δήλωση της κυρίας ε, στον κατά της εθνικοποίησης της Ρεψόλ από την κυβέρνηση της Αργεντινής. Αυτό όμως ε, είπατε ότι θα πρέπει να συγχαίει οικονομικά με τα εθνικά συμφέροντα. Ελπίζω την ίδια δυναμικότητα και την ίδια ζέση να, να δείξετε και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των 15 Κούρδων που αυτή τη στιγμή πραγματοποιούν απεργία πείνα στο Στρασβούργο ω ένδειξη διαμαρτυρία. Σε ό,τι αφορά τη Δυτική Σαχάρα, ε, την κατάσταση στη Λωρίδα τη Γάζα και τα κατεχόμενα και σε πάρα πολλέ άλλε περιπτώσει ε, που είναι πονίδιστες ε, και δεν περιποιούν καθόλου τιμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στους Ευρωπαίους πολίτες. Ο κύριος Χόιτ στην εξαιρετική του έκθεση μιλάει για τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών και τους μηχανισμούς συμμετοχής στις διαπραγματεύσεις για τις εμπορικές διαπραγματεύσεις και τις, την ανάγκη διαβουλεύσεων και ενημέρωσης πριν τη σύναψη συμφωνιών με τους αυτόχθονες πληθυσμούς. Ευχαριστώ. Ο κύριος Φερέιρα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση που ε, σπέβδει να δώσει κηρύγματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, σε όλο τον κόσμο ε, διαπιστώνει παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων εντός Τη επικράτεια τη δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλιση, προστασία κατά τη ανεργία, δίκαιο και αξιοπρεπή μισθό, δικαίωμα στη διατροφή, στην υγεία, στη δωρεάν εκπαίδευση. Και αυτά είναι ανθρώπινα δικαιώματα που περιλαμβάνονται στην οικουμενική διαχείριση, αλλά όλα αυτά στην οικονομική, οικουμενική, οικουμενική διακήρυξη. Αλλά δυστυχώ στην Πορτογαλία, στην Ελλάδα και σε άλλε χώρε πέφτουν θύματα στο βωμό των ε, σχεδίων λιτότητα, των μνημονίων και τις ε, προσπάθειες εξηγήσεις των οικονομικών. Θα πρέπει ε, να μην ε, υπερασπίζουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά εις βάρος των δικαιωμάτων των εθνών και των πολιτών, καταπατώντας τους στοιχειώδες κανόνες της δημοκρατίας. Τα ανθρώπινα δικαιώματα χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο ως πρόσχημα για την επέμβαση στα εσωτερικά χωρών, καταστρατηγώντας το πνεύμα και το γράμμα των Ηνωμένων Εθνών και των συμβάσεων του ΟΗΕ. Νομίζω ότι είναι πολύ συσταλτική και επιλεκτική η ερμηνεία που κάνουμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει η Λεδιάστον. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Όπως αναφέρθηκε στη συζήτηση, είναι μεγάλο το πεδίο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των οικουμενικών ιδιαίτερα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και τη οικουμενικότητα, του οικουμενικού χαρακτήρα του. Εγώ θα αναφερθώ σε ορισμένα από αυτά. Θα ήθελα καταρχήν να εκφράσω την ιδιαίτερη μου ικανοποίηση για την αποφυλάξη των κυρίων Σενέκο και Μποντερέγκο στη Λευκορωσία. Χαιρόμαστε για την αποφυλάξη των δύο πολιτικών κρατουμένων και νομίζω ότι ίσως δίνει μια ευκαιρία και στη Λευκορωσία, δείχνει τη βιγμή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το σθένος της και την αποφασιστικότητά της. Και δείχνει επίσης ότι η Ένωση, η σύμπνοια στα θέματα αυτά είναι πολύ σημαντική γιατί δημιουργεί την ισχύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το θέμα της πίστης, της δοξασίας, της θρησκευτικής λατρείας, η δυνατότητα να μπορεί κανείς ε, να ασκήσει το δικαίωμα λατρείας, ε, είτε πιστεύει είτε όχι σε μια θρησκεία είτε ανήκει σε μια θρησκεία. Είμαι υπέρ αυτών των δικαιωμάτων και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την συμπερίληψη αυτών των δικαιωμάτων ε, στις μελέτε που κάνουμε για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Γι' αυτό και στην ετήσια έκθεση αφιερώνουμε ένα ειδικό κεφάλαιο στο θέμα της ανεξιθρησκεία. Δίνεται ιδιαίτερη σημασία και στον τομέα αυτό τη ελευθερία, δοξασία ε, και θρησκευτική λατρείας. Ε, φυσικά μας ε, θορυβή κατάσταση στην Αίγυπτο και παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Ο κύριος Ντόνσκης μίλησε και για τις ε, πολύ πιο εκλεπτισμένες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την πρόκληση που αντιμετωπίζουμε ε, να αντιμετωπίσουμε όχι μόνο κατάφορες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων όπως είναι η θανατική καταδίκη. Ζητούμε κατάργηση της θανατικής ποινής. Αυτό είναι σημαντικό και θεμελιώδες τμήμα της προσπάθειάς μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά να ε, δούμε και πώς ε, στερούνται ορισμένοι των δικαιωμάτων τους ή εμποδίζονται από την άσκηση των δικαιωμάτων τους, που είναι μια πιο εκλεπτισμένη μορφή παραβίασης. Επίσης, η έλλειψη αξιοπρέπειας, η έλλειψη σεβασμού ε, συνιστούν παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το μήνυμα για την Αργεντινή δεν είχε καμία σχέση με τη συζήτηση ε, Απλώ ε, με ρώτησε ο κύριο Αλαφράγκα, θα μπορούσα να πω κάτι πριν την έναρξη τη συζήτηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν συνδυάζεται η συζήτηση αυτή με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Συμφωνώ με την ε, αποτρόπια κατάσταση που επικρατεί στη Γουινέα Μπισάου. Και πριν το πραξικόπημα τη προηγούμενη πέμπτη, ήδη είχα ε, εκφωνήσει δήλωση και ζήτησα σεβασμό από τις αντιπαλόμενες πλευρές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ζήτησα ε, απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων και μάλιστα ανεστάλλει βοήθεια προς τη Γουινέα Μπισάο μέχρι ότου διορθωθεί η κατάσταση και συνεχίζουμε την άμεση υποστήριξή μας προς το λαό. Δεν πρόκειται να υποστηρίξουμε μια παράνομη κυβέρνηση, μια πραξικοπηματική κυβέρνηση. Μην νομίζετε ότι προσπάθησα να εμπλέξω τα δύο θέματα. Η Αργεντινή ήταν ένα ξεχωριστό ζήτημα από την συζήτηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και προηγείται τη συζήτηση αυτή. Συμφωνώ με όσους ζήτησαν το διορισμό του ειδικού εντεταλμένου για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όπως ξέρετε αυτή τη στιγμή επεξεργαζόμαστε την εντολή για τον ειδικό εντεταλμένο και να ζητούμε κάποιον που θα χαρακτηρίζεται από ακαιρεότητα και θα έχει και σημαντικέ δεξιότητε και προσόντα και ικανότητε. Γιατί θα είναι πολύ σημαντικό ο ρόλο και θα πρέπει ο ειδικό αυτό εντεταλμένο να έχει συνεργασία και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα συνεχιστεί λοιπόν η συζήτηση για το θέμα αυτό. Με ιδιαίτερη χαρά διαπίστωσα ότι πολλοί αναφέρθηκαν στο θέμα των δικαιωμάτων των γυναικών και τη σπουδαιότητα που έχει η υποστήριξη των γυναικών, ιδιαίτερα εκείνων που διαβιούν σε ακραίες συνθήκες τρόμου και φρίκης και φυσικά να προσπαθούμε να τις αναμίξουμε στην οικονομική και κοινωνική ζωή των χωρών στις οποίες διαμένουν. Γνωρίζουμε ότι οι γυναίκες ε, όπου συμμετέχουν στις κοινωνίες ε, εμπλουτίζουν τις κοινωνίες αυτές και από κοινωνική, από οικονομική αλλά και από πολιτική άποψη. Και το θέμα των ε, αναγκαστικών γάμων δυστυχώς μαστίζει πολλές χώρες. Όταν ήμουν ε, Υπουργό Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην πατρίδα μου, προήγαγα ε, νομοθεσία για την ε, απαγόρευση τέτοιων αναγκαστικών γάμων. Είναι ένα ζήτημα που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε σοβαρά όπου και αν εμφανίζεται. Κυρία Λάτφορτ, ξέρετε ότι ασχολούμαστε με το θέμα αυτό και ξέρετε ότι με προβληματίζει ιδιαίτερα η ισχύ τη θανατικής ποινής. Ήδη φέτος στο Ιράν είχαμε 100 εκτελέσεις ε, πρωτοστατήσατε με τις προτάσεις σας ε, ε, για το θέμα αυτό και μάλιστα ασκούμε πίεση στα κράτη-μέλη και ζητούμε τη βοήθεια των ευρωβουλευτών για να ε, επανεγκαταστήσουμε όλο και περισσότερους. Ε, ε, ξέρω κύριε Στίβενσον ότι σας ενδιαφέρει αυτό το θέμα του στρατοπέδου, του καταβλισμού ΑΣΡΑΦ και υπάρχει και οικονομική υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να βελτιωθεί η κατάσταση. Και μάλιστα όσο περισσότερη υποστήριξη δώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τόσο πιο εύκολα θα προωθήσουμε το θέμα. Πάντω, Σα διαβεβαιώ ότι και εμά μα απασχολεί ιδιαίτερα το θέμα και μεριμνούμε γι' αυτό. Σε ό,τι αφορά την Νότια Αφρική, ναι, συμφωνήσαμε για διάλογο για ανθρώπινα δικαιώματα με την Νότιο Αφρική. Εκεί θα θίξουμε πολλά και διάφορα ζητήματα και συμφωνώ με την κυρία Γκόλτμαν για τη σημασία επαφής και συνάντησης με ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό επιδιώκω σε κάθε χώρα που επισκέπτομαι. Και θέλω να έχω ανταλλαγή απόψεων μαζί τους για να ακούω ε, αυτόπτες μάρτυρες της κατάστασης ε, και ζητώ ενημέρωση για την καθημερινότητα αυτών των ανθρώπων. Και φυσικό είμαι υπέρ ε, και των δικαιωμάτων των ΛΟΑΔ, των λεσβιών, ομοφιλοφίλων, αφιφιλοφίλων και διαφιλικών. Θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να υπερασπίσουμε και τα δικά του δικαιώματα, που και αυτά εμπίπτουν στα οικουμενικά ανθρώπινα δικαιώματα. Μίλησα προηγουμένω ε, για την ανάγκη να έχουμε την ένταξη και όχι τον αποκλεισμό. Και τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι δείκτης για την συνεργασία μας με τρίτες χώρες. Πολύ συχνά συνεργαζόμαστε με εκπροσώπους των χωρών προκειμένου να βελτιώσουμε τη θέση της κοινωνίας των πολιτών, ενώ ταυτόχρονα προσπαθούμε να απομονώσουμε και να ασκήσουμε πίεση στις κυβερνήσεις τους. Δεν θέλουμε να εγκαταλείψουμε στη μοίρα τους ανθρώπους που φροντίζουν να ασκήσουν και να υπερασπίσουν τα δικαιώματά τους. Δεν θα αφιστούμε προ... προσπαθειών να τους βοηθήσουμε. Θα πρέπει να συνδυάσουμε λοιπόν την στήριξη του λαού με την απομόνωση των αυταρχικών κυβερνήσεων. Μόνο έτσι θα βελτιώσουμε την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και ένα πιο γραφειοκρατικό ζήτημα, το benchmarking, την ε, συγκριτική την συγκριτική αξιολόγηση και την μεθοδολογία για να αποτιμήσουμε τις επιδόσεις των διαφόρων χωρών στα ανθρώπινα δικαιώματα. Βέβαια, πολύ δρόμο έχουμε να διανύσουμε ακόμη, αλλά νομίζω ότι η αφετηρία μας είναι πολύ καλή. Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμότατα τον εισηγητή για το έργο του σε αυτή την πολύ σημαντική έκθεση. Γνωρίζω ότι είναι δεδομένη η προσωπική σας ε, δέσμευση και στράτευση για το θέμα αυτό και θα ήθελα να αποτίσω φόρο τιμής σε αυτήν ακριβώς τη στράτευση. Ευχαριστώ την Βαρόνη. Το λόγο έχει ο κύριος Χαουίτ για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ γιατί η συμβολή σας είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίσουμε το ρόλο του ειδικού εντεταλμένου, το θέμα της λογοδοσίας, στις ε, δηλώσεις των θεσμικών οργάνων. Ε, πολύ σημαντικό είναι αυτό που αναφέρθηκε για τους αναγκαστικούς γάμους, τη συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη, την προσέγγιση της θανατικής καταδίκης, ποινής κλπ. Ευχαριστώ για όλα τα καλά λόγια που άκουσα και από τους Σκιώδης ε, στηρίζω την ε, πρόταση του κυρίου Γκρίψε η οποία θα ε, ζητήσω να ενσωματωθεί. Επίσης ο κύριος Μπρόκο και η κύριε Μπρόκ, Ματέρα, Καρλ από την ομάδα ΕΛΚΑ έδειξαν ότι μπορούμε να είμαστε επικοδομητικοί και να έχουμε μια διακομματική συνένεση. Σε ό,τι αφορά τώρα την ε, προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση. Αυτό έχει συζητηθεί και εδώ και στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης. Είναι σαφές ότι είναι κατά το Ηνωμένο Βασίλειο ε, ε Βαρόνι Λάντφορντ και ε, υπάρχει η ελπίδα να αλλάξει αυτό αργότερα κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Θα δούμε. Ε, σε ό,τι αφορά τώρα τα διπλά μέτρα και σταθμά. Βεβαίως αυτό είναι σημαντικό και για τη συζήτησή μας. Ε, Στη Νότια Αφρική καταδικάζουμε δολοφονίες ε, λευκών και μαύρων. Ε, ναι, έγινε αναφορά στην Αργεντινή, όχι στην Κολομβία και εκφράστηκαν ορισμένες ανησυχίες από τους κυρίους Πόσελ και άλλους σε σχέση με την εξέλιξη μετά την Αραβική άνοιξη. Ε, σημαντικό είναι και στην περιοχή αυτή αλλά και σε όλο τον κόσμο να καταδικάσουμε ε, καταχρηστικές πρακτικές ε, σε ό,τι αφορά ε, το πρόβλημα της ομοφιλοφιλίας ε, και τα προβλήματα λεσβιών και άλλων τέτοιων ομάδων ε, βεβαίως θα πρέπει να αλλάξουν οι πρακτικές που προβλέπουν ότι η ομοφιλοφιλία είναι ασθένεια. Υποστηρίζω τις σχετικές τροπολογίες. Επίσης τα νούμερα που μας έδωσε η κυρία Άστον είναι σωστά. 28 εισηγητές για τα ανθρώπινα δικαιώματα υπήρξαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά τι πρώτε άμεσες εκλογές Ε, αυτό είναι αλήθεια και καλό είναι να συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. τέλος θα ευχαριστώ πολύ που μου ανατέθηκε η έκθεση αυτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κλείνει εδώ η συζήτηση. Η ψηφοφορία θα γίνει αύριο στις 11.30. Τώρα στην ημερήσια διάταξη έχουμε τη δήλωση της ύπατης εκπροσώπου